Okay, ladies we can Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αν και εφόσον το επιθυμείτε και η τεχνική ε, νομίζω ότι είναι εντάξει, είναι στη θέση της η τεχνολογία χρειάζεται λίγο χρόνο αλλά τελικά λειτουργεί. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Έχετε την, ε, το σχέδιο ημερήσιας ε, διάταξης, ε, την έχετε στο φακελό σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση που θέλετε να κάνετε. Υπάρχει όμως και μια μικρή αλλαγή για το σημείο 8, το οποίο έχει αντικατασταθεί από την παρουσίαση από την Κομισιό το τι συμβαίνει τώρα, μας, θα μας παρουσιάσει η Κομισιόν τι συμβαίνει τώρα και το τι πρόκειται να συμβεί στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου. Αυτό είναι η αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Δεν έχω ανακοίνωση. Okay. Then we can start. Εφόσον δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του Connecting Europe Facility και ο τίτλος δύσκολος είναι ήδη. Και έχουμε και την, ε, ε, την παρουσίαση των ε, τομεακών επιπτώσεων των διευρωπαϊκών δικτύων, των ομολόγων έργου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις υποδομές των τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα μας πολύ σημαντικό και γι' αυτό έχουμε και πολλούς εκπροσώπους της Κομισιόν σήμερα εδώ που θα κάνουν μια κοινή παρουσίαση και αν συμφωνείτε ε, θα δώσουμε για την, ε, τις διαφορετικές πτυχές των, ε, της παρουσίασης κάποια χρονικό όριο, να καλωσορίσω τους παρισταμένους, τους προσκεκλημένου μας και θα ξεκινήσουμε πρώτα με ποια σειρά. Εσείς θα ξεκινήσετε πρώτα. Ωραία. Ευχαριστώ, πολύ για την ευκαιρία που δίνεται στην Κομισιόν να παρουσιάσει το CEF, το Connecting Europe Facility. Θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε συντονισμένα και ολοκληρωμένα, διότι ούτως ή άλλως και το εργαλείο αυτό είναι συντονισμένο. Θα παρουσιάσουμε καταρχάς το υπόβαθρο, την μηχανική με την οποία λειτουργεί, το όλο σύστημα και μετά θα σας παρουσιάσουμε την ενέργεια και την διάσταση της κοινωνίας πληροφορικής. Και μετά θα αναφερθούμε και στα καινοτόμα ε, τις καινοτόμες ε, δυνατότητες χρηματοδότησης. Λοιπόν, το CEF είναι ένα κομμάτι ενός συνολικού πακέτου, το οποίο υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο από την Κομισιό μέσα στα πλαίσια του οικονομικού του χρηματοδοτικού πλαισίου, αλλά και μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας ολοκλήρωσης της ε, εσωτερικής αγοράς. Μιλάμε για ενοποίηση, για ολοκλήρωση, για συνεργασία για κοινοτική προστιθέμενη αξία. Εξετάζουμε τρεις τομείς, κοινωνία πληροφορικής, ενέργεια και μεταφορές. Εξετάζουμε συνεργασίες και ολοκλήρωση ανάμεσα στον, στα πλαίσια προγραμματισμού και για τις ε, κατευθύνες γραμμές TEN. Επίσης εξετάζουμε την συνεργασία ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση σε διαφορετικό επίπεδο βέβαια, σε όλους τους τομείς που μας απασχολούν. Επίσης εντοπίσαμε και προσπαθήσαμε να, να υπογραμμίσουμε την κοινοτική προστιθέμενη αξία σε συνεργασία και με τις προσπάθειες που καταβάλει ο βιομηχανικός τομέας και τα κράτη-μέλη και πέραν τούτου όμως, με τη συνεργασία που έχουμε με τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, καταβάλαμε περαιτέρω προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το CEF να προσφέρει και προστιθέμενη αξία και σε άλλα εργαλεία σε κοινοτικό επίπεδο, παραδείγματο χάρη κάποια ε, ταμεία ενέργειας ε, με τον ορίζοντα του 2020, αλλά και μετά διάφορα εργαλεία που έχουμε στη διαθεσή μας για τις εξωτερικές διαστάσεις της κοινοτικής πολιτικής. Επομένω, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από πλευρά της Κομισιό, που εκπροσωπείται και φυσικά Φυσικά σε αυτό το βήμα τέσσερις εκπρόσωποι, μάλλον εκπρόσωποι τεσσάρων γενικών διευθύνσεων που είναι εδώ, ΕΚΦΙΝ, ΕΝΕΡ, ΙΝΦΟ και εμείς. Από, και εμείς από την... Τώρα θα κάνουμε μια, υπάρχει και μια γραπτή παρουσίαση την οποία μπορούμε να σας δώσουμε αλλά τέλος πάντων θα την παρουσιάσουμε πάρα πολύ σύντομα διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενέργεια και η κοινωνία της πληροφορικής αλλά για να επανέλθω στα βασικά στοιχεία αυτού του instrument, αυτού του εργαλείου ποια είναι η προστιθέμενη κοινωτική αξία και να ξέρουμε ότι αυτό το εργαλείο είναι εδώ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των υποδομών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εσωτερική αλλά και για τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, αλλά και για την κοινοτική υποδομή που στηρίζει την ανταγωνιστικότητά μα και όσον αφορά την γενική οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους τρεις τομείς, διότι όλοι αυτοί οι τομείς μας βοηθάνε να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα καθενός από τους τρεις τομείς όπου θα βρείτε ότι στην κοινωνία της προφορική, στις μεταφορές και στην ενέργεια θα δείτε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη που παραμένουν ηγέτες, παγκόσμιοι ηγέτες στις υπηρεσίες, στον εξοπλισμό και στα συστήματα. Επομένως αυτό το CEF, αν θέλετε, αυτό το εργαλείο που ενώνει την Ευρώπη, θα υποστηρίξει γενικότερα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στους τρεις τομείς. Τώρα, εν συντομία, να σας πω ποιε είναι οι, ποιες είναι οι επενδύσεις και οι δείκτες. Ε, στις κατευθυντήριες γραμμές που υποστηρίζουν, αν θέλετε, που είναι ένα παράρτημα ε, του CEF, αλλά και στα παραρτήματα, η Κομισιό έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε να εντοπίσουμε ποια συγκεκριμένα, ποιες συγκεκριμένες είναι οι επενδύσεις ε, σε τομείς και σε project που έχουν την μέγιστη ε, κοινοτική προστιθέμενη αξία. Αλλά όλα αυτά βέβαια και σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε για τις επενδύσεις. 50 δις εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011 και υπάρχει μια κατανομή σε τρεις τομείς είναι διαφορετικά τα ποσά βέβαια και αυτό αντικατοπτρίζει όχι, όσο τόσο, όχι τόσο τις ανάγκες επένδυσης ε, και τις κατευθύνες γραμμές αλλά την ανάγκη ε, για, περαιτέρω, για συμπληρωματική κοινοτική χρηματοδότηση σε σχέση με την εθνική χρηματοδότηση. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό το εργαλείο ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε ολοκληρωμένα γιατί η αποτελεσματικότητα είναι το κύριο στοιχείο Επίσης θα πρέπει να κάνουμε και την επιλογή, να έχουμε ένα πιο κεντρικό σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων που δίδονται, ε, γιατί δεν είναι η Κομισιόν που θα διαχειρίζεται το Ταμείο, αλλά η Κομισιόν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο βέβαια και με τα κράτη-μέλη και, με βάση, και με, σε συνεργασία με την Επιτροπή που θα δημιουργηθεί, ε, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα project τα οποία έχουν την μέγιστη κοινωτική προστιθέμενη αξία. Και υπάρχει και ολόκληρο σύστημα για, τον, για την προκήρυξη των διαγωνισμών κτλ. που ακριβώς αυτά τα κριτήρια ακολουθεί. Προσπαθούμε να αποφύγουμε Υπάρχουν μα βέβαια και, κάποιες, και κάποιοι ενδιάμεσοι, όπως παραδείγματος χάρη το, ε, η Ευρωπαϊκή ε, τράπεζα Επενδύσεων, ε, αλλά στους, στις, θα τα δούμε αυτά αργότερα, αλλά στις μεταφορές ε, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα διοικητικά προσπαθούμε να τα δώσουμε έξω. Υπάρχει, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιες agencies, κάποιοι οργανισμοί που θα αναλάβουν τη διαχείριση του εργαλείου αυτού μετά το 2014. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο. Επίσης ε, εξετάζουμε πώς θα γίνει αυτό στους άλλους δύο τομείς, στην ενέργεια και στην κοινωνία της προφορικής. Και η εφαρμογή του project επιτόπου βέβαια, τα συμβόλαια, οι προμήθειες, όλα αυτά παραμένουν ευθύνη των κρατών μελών και ε, των δικαιούχων, αν θέλετε, που είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα, μέσω ενός ε, ενιαίου κανονισμού και μέσω ενός ε, ενιαίου μηχανισμού λειτουργίας ε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο βαθμό ευελιξίας και ανάμεσα στους τομείς υπάρχει και μια midterm review η οποία προβλέπεται και οι τρεις γενικές διευθύνσεις πιστεύουν ότι τα ποσά όλα αυτά είναι λογικά και μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Επομένως, πιστεύουμε ότι αυτοί οι τρεις τομείς θα ξεκινήσουν αποτελεσματικά ευθύ εξ αρχής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και κάποιο περιθώριο ευελιξίας, εάν παραστεί ανάγκη. Επίσης υπάρχουν και εργαλεία, καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν την έχουμε όμως καταγράψει, αν θέλετε, ακόμα. Ε, όμως θα το καθορίζουμε σε αιτήσια βάση όσο προχωράει η εφαρμογή του CEF. Και όλα αυτά βέβαια θα είναι σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα δημοσιονομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, περνάμε στους δύο τομείς που ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας, η ενέργεια καταρχάς και δίνω το λόγο στην συνάδελφο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για τον κλάδο της ενέργειας, όπως ξέρετε και εσείς, ε, είχε ανατείλει μια νέα εποχή όπου χρειάζεται επίγουσα δράση και βεβαίως και μια νέα προσέγγιση στην πολιτική που χαράσουμε. Πρέπει να κλείσουμε καταρχήν το θέμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και να ενώσουμε τα ενεργειακά, τις ενεργειακές νήσους όπως τις ονομάζουμε με το κέντρο της ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2015 όπως αποφάσισαν οι αρχαίοι κρατών και κυβερνήσαν πρόσφατα. Αυτό βεβαίως αφορά και τις χώρες της Βαλτικής αλλά και την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ελλάδα. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια και αέριο οποιαδήποτε στιγμή χρειάζονται σε καλές τιμές. Κάθε χρόνο όσο μπαίνει ο χειμώνας, ο κίνδυνος για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό επανακάμπτει, άρα λοιπόν και εδώ επίγει να δράσουμε. Είναι γνωστή η το, είναι γνωστό το πόσο ευαίσθητο θέμα είναι το φυσικό αέριο στις χώρες της ε, πιο ανατολικές και κεντρικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι χώρες αυτές ε, καταρχήν δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και σε θαλάσσιες μεταφορές αερίου, αλλά επίσης εξαρτώνται από έναν και μοναδικό αγωγό φυσικού αερίου. Για την ηλεκτρική ανέργεια θα θυμόσαστε πως το 2006 15 εκατομμύρια πολίτες από τη Γερμανία μέχρι και τη Βόρεια Ιταλία έμειναν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια γιατί το δίκτυό μας δεν ήταν αρκετά ευέλικτο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια, ένα μικρό blackout. Για να επιτύχουμε λοιπόν τους στόχους αυτούς για τον ανεφοδιασμό που επίγουν όπως σας είπα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στη ζήτηση και αυτό βεβαίως προϋποθέτει ένα ευέλικτο δίκτυο. Η βιωσιμότητα, η ΑΠΕ, η Ευρώπη αποφάσισε μέχρι το 2020 να εφοδιάζεται με 20% ενέργεια από ΑΠΕ. Έχουμε συμφωνήσει δε να μέχρι το 2050 να έχουμε ε, απελευθερώσει την εξάρτηση από τα άνθρακούχα ε, κατά 85-90%. Which again requires interconnected networks and flexible networks. Θέλουμε λοιπόν διαλειτουργικά δίκτυα τα οποία θα είναι όπως σας είπα ευέλικτα στις χώρες της Βόρειας Θάλασσας Και βεβαίως υπάρχει και η παραγωγή ενέργειας από η παλιροϊκή ενέργεια και η αιωλική ενέργεια. Δυστυχώς όμως αυτό δυσκολεύει τις χώρες οι οποίες είναι μακριά από τα παράλια και τις ακτές. Χρειάζεται λοιπόν να βασιστούμε στην ηλιακή ενέργεια, ηλιακή ενέργεια η οποία στα κράτη της Μεσογείου είναι άπλετη. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και ε, τις διακυμάνσεις που έχουμε ε, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και διασυνδέσεις αλλά και backup το οποίο προσφέρει η ευέλικτη διασύνδεση με αέριο κτλ. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα προσφέρουν το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μοχλευθούν οι απαραίτητες επενδύσεις εμπρό έτσι ώστε να επιβιώσει ο κλάδος αυτός της βιομηχανίας μας. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ορίσει 12 διαδρόμους προτεραιότητας και όχι μόνο διαδρόμους αλλά και κλάδους προτεραιότητας. Καλύπτουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Βλέπετε στο χάρτη που βρίσκονται. Εννέα λοιπόν γεωγραφικοί διάδρομοι και τρεις θεματικές περιοχές ε, που έχουν τα ευφυή δίκτυα, για παράδειγμα τα δίκτυα ε, διοξιδίου του άνθρακα και τις, ε, τους αυτοκινητοδρόμους της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές, για τις υποδομές, παρουσιάζουν κάποιους μηχανισμούς που θα μετατρέψουν αυτούς τους διαδρόμους και χώρους σε συγκεκριμένα έργα ε, στο περιφερειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τεχνικά κριτήρια τα οποία θα απηχούν τους στόχους που έχει η πολιτική μας. Η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι ευέλικτη και θα επαναλαμβάνεται η εξετασία της κάθε δύο χρόνια έτσι ώστε ε, να λαμβάνονται υπόψη και τα όσα θα πούνε οι παίκτες, οι μεγάλοι οικονομικοί παίκτες ε, του κλάδου όσον αφορά το δυναμικό και τις δυνατότητες τις τεχνικές δυνατότητες που εμφανίζονται. Έχουμε λοιπόν κάποια εργαλεία που θα επιτρέψουν την εμπρόθεσμη εφαρμογή και επαναλαμβάνω θα μοχλεύσουν το ιδιωτικό κεφάλαιο που χρειάζεται. Το πιο βασικό είναι πως η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την επιτάχυνση της αδειοδότησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων. Είδαμε στην πράξη πως χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια και στις χειρότερες περιπτώσεις μέχρι και 30 χρόνια έτσι ώστε να έχει κανείς να λάβει άδεια για να χτίσει δίκτυο. Δεν έχουμε 10 χρόνια μέχρι το 2020, είμαστε στο 2011, οπότε πήγε. Stop shop. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξυπηρέτηση της ενιαίας θηρίδας στα κράτη-μέλη με, μια, με ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών μέχρι να χορηγηθεί άδεια. Europe, we are very proud of our high environmental standards and therefore the proposal also... Να μπορούμε λοιπόν να εισάγουμε νέες υποχρεώσεις για, τους, για όσους προωθούν τις ε, νέες αυτές ε, διασυνδέσεις, να εμπλέξουμε πολύ περισσότερο τους πολίτες, ακόμη και άλλους παίκτες οικονομικούς σε όλη τη διαδικασία και να παράσχουμε και, την, και τις καλύτερες ποιοτικές πληροφορίες για όλα αυτά τα προγράμματα σε όσους βεβαίως ενδιαφέρονται και βεβαίως θα δούμε και πώς θα εξασφαλίσουμε και την ε, διάσταση την ε, ποιοτική ε, στους από πλευράς αναδόχων. Βασιζόμαστε λοιπόν σε τιμολόγηση με τέλη τα οποία θα καταβάλουν οι χρήστες και στην πρότασή μας έχουμε ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο επεκτείνοντας την αρχή ο, καταναλωτής ε, πληρώνει λίγο πιο πολύ. Έτσι λοιπόν όποιος ωφελείται από αυτά θα πληρώνει το αντίτιμο. Οι επενδύσεις στη μία χώρα ε, πολλές φορές δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους πολίτες κάποιας άλλης χώρας. Σήμερα είναι αδύνατο να ζητήσουμε από τη γείτονα χώρα να συνεισφέρει στην χώρα που επενδύνει, παρόλο που μπορεί να δρέπει τα πλεονεκτήματα αυτής της εθνικής επένδυσης. Θα κάνουμε λοιπόν μία κατανομή κόστους για όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια όπου ε, το κόστος και τα ωφέλη έχουν κατανεμηθεί με ασύμετρο τόπο. Και για να συμπληρώσουμε αυτό το πακέτο και να εξασφαλίσουμε πως τα project αυτά, θα, τα έργα αυτά θα έχουν και κάποια μη εμπορικά πλεονεκτήματα, ωφέλη, δηλαδή αλληλεγγύη, ε, διασύνδεση της Ευρώπης κτλ. Ο μηχανισμός μας θα συμπληρώσει το ε, ε, ρυθμιστικό πλαίσιο όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Για την ενέργεια λοιπόν δεν έχω κάτι ακόμα να προσθέσω. Θα ήθελα να... Να σας κάνω εγώ μια μικρή εισαγωγή για το τρίτο τμήμα του CEF που έχει να κάνει με τις υποδομές στην Ευρώπη του μέλλοντος. Θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή είναι πολύ παθιασμένη έτσι ώστε όλος, όλοι οι Ευρωπαίοι να περάσουν σε μια ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι κομμάτι και της ψηφιακής ατζέντα που έχει αποτελέσει σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το CEF είναι ένα κομμάτι των προθέσεων που έχουμε ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Το CEF στο, στο διαδίκτυο βασίζεται σε δύο πυλώνες. Όποιους ε, έχουν δει τον ε, πίνακα των ε, βαθμολογιών που έχουμε, των επιτυχιών μας, βλέπετε ότι υπάρχουν δύο πτυχές που χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία είναι να διευκολύνουμε την ψηφιακή πραγματικότητα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 Ε, και των, ε, της διευρυζωνικής σύνδεσης και των υποδομών. Η διευρυζωνική σύνδεση βεβαίως θα μας βοηθήσει να έχουμε γρήγορο ίντερνετ και αυτό ως πολίτες και ως καταναλωτές αλλά και ως επιχειρήσεις μπορούμε να ε, το χρησιμοποιήσουμε και βεβαίως στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Ο άλλος πυλώνας της πρότασης έχει να κάνει με την διαθεσιμότητα των δημοσίων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες είναι περισσότερες online στις περισσότερες χώρες. Η πρόθεσή μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Επίτροπος, ε, όπως είπε ο Επίτροπος Μεταφορών, να μην καταλήξουμε σε μια ε, ενιαία αγορά που να είναι κατακριματισμένη και να μην αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να έχουν μια ε, ενιαία πλατφόρμα που θα μπορέσει να τις καταστήσει πραγματικά ευρωπαϊκές. Η ευρωπαϊκή ατζέντα έχει φιλόδοξους στόχους για το τι σημαίνει η αποδεκτή, τι σημαίνει αποδεκτή συνδεσιμότητα. Έχουμε προτείνει όλοι οι Ευρωπαίοι μέχρι το 2020 να έχουν πρόσβαση σε ε, ταχύτητες 30 MB το δευτερόλεπτο. Ε, τα μισά νοικοκυριά της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ε, τουλάχιστον 100 MB το δευτερόλεπτο τέτοιες ταχύτητες. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπτυξη της ε, διαβριζονικότητας, ε, που είναι μια διαδικασία που οποία ε, της οποίας ηγείται κυρίω ο ιδιωτικό τομέα και βεβαίω περιέχει και πολλού κινδύνου. Θεωρούμε ότι η δική μα στήριξη θα πρέπει να γίνει μέσω τη υποστήριξη των δυνάμεων τη αγορά, να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να ξεφύγουν από το πρόβλημα των επενδύσεων. Δυστυχώ, η ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί μια προσφορά για λίγου για λίγους Ευρωπαίους. Ε, σίγουρα αυτοί θα, είναι αρκετά, θα έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα και θα ζουν και σε πύκνα κατοικημένες περιοχές της Ευρώπης. Η εμπορική προσφορά για τα επόμενα χρόνια, χωρίς παρέμβαση, δεν θα προχωρήσει πέρα από αυτά τα δεδομένα. Οπότε θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος που μίλησε για τα δημοσιονομικά εργαλεία, αλλά θεωρώ και εγώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πρόκλησης μπορεί να αντιμετωπιστεί δίνοντας το σωστό ε, ρυθμιστικό περιβάλλον πάνω στο οποίο βεβαίως δουλεύουμε και τα χρηματοοικονομικά ε, εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτής της επένδυσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν υποδομές ε, για τις τηλεπικοινωνίες. Και αυτό θα είναι ένα μακροπρόθεσμο, μακρόπνο σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη. Τώρα, να δούμε τις λεπτομέρειες των online δημοσίων υπηρεσιών. Γιατί πρέπει να είναι ευρωπαϊκές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, η καταγραφή ενός παιδιού σε ένα μητρό ή ενός αυτοκινήτου από μια χώρα σε άλλη. Είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σήμερα, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και πολύ δαπανηρό και αυτό βεβαίω το αναλαμβάνει ο καταναλωτή ή η επιχείρηση. Αυτοί πρέπει να ε, ασχοληθούν με όλα τα διοικητικά έγγραφα, να μεταφραστούν στι σωστέ γλώσσες. Δεν υπάρχει ε, ανάγκη τα συστήματα να μην είναι ε, διασυνδεδεμένα. Στο σχετικό πρόγραμμα που έχει υπάρξει αποδείξαμε ότι η διαλειτουργικότητα πολλών από αυτές τις υπηρεσίες είναι δυνατόν να γίνει εφικτή. Στο ΣΥΕΦ θα θέλαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα προς τα εμπρός, το επόμενο λογικό βήμα, που είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, ώστε να κάνουν και αυτά με τη σειρά τους το δικό τους βήμα προς τα εμπρός, σε ό,τι αφορά τις δικές τους εθνικές δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ευρώπη, στη σωστή γλώσσα, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω γραφειοκρατία και χωρίς επιπλέον κόστος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για να γίνει πολύ πιο εύκολη η χρήση όλων αυτών από τους Ευρωπαίους, αλλά και για να μειωθεί το κόστος των δραστηριοτήτων των επιχειρησιακών στην Ευρώπη γιατί μιλάμε για, πολύ, ε, για εταιρείες υψηλής ε, τεχνολογίας που ε, μπορεί να περάσουν και 18 μήνες για να θέλουν, για να σκεφτούν ότι μπορεί να ξεκινήσουν μια τέτοια επένδυση για να επιβιώσουν στην οικονομική αγορά. Και είναι σημαντικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να, να γίνουν ευρωπαϊκές και να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ευρώπη. Η διαφορά του να έχεις ή να μην έχεις πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες online στο, με το σωστό τρόπο και στη σωστή γλώσσα για να μειώσουμε το κόστος στην ε, Ευρώπη βεβαίως είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ως παράδειγμα του τι σκεφτόμαστε γι' αυτό, θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι την εντύπωση ενός σύννεφου αντί για διασυνοριακή σύνδεση. Ξέρετε ότι η Κομισιόν ήδη έχει εισάγει, έχει δημιουργήσει μάλλον το πόρταλ Europeana, το οποίο έχει, για το, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και το οποίο ψηφιοποιείται από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι το σημείο εισόδου ε, εξασφαλίσαμε ότι μπορούμε όλοι να το χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικού σκοπούς, για επιχειρησιακούς σκοπούς και δεν έχει αλλάξει ο κανόνα, ανάλογα με την, δεν αλλάζουν οι κανόνες ανάλογα με τη, με τη χώρα. Και οι δημόσιοι, όσες λοιπόν οι δημόσιε υπηρεσίες είναι δημόσιες, η δική μας βασική παρέμβαση θα είναι μέσω επιδοτήσεων και συμβάσεων. αλλά η αμοιβαία ενίσχυση, η υποστήριξη αυτής της πρότασης έχει να κάνει με το ότι η χρήση των φυσικών δικτύων θα αυξήσει και θα βελτιώσει τις, ε, τις ε, επιχειρήσεις. Ενώ η ασφάλεια που θα έχουν αυτές οι φυσικές υποδομές θα μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να, κάνουν, να καταστήσουν διαθέσιμες τις online ε, δημόσιες υπηρεσίες τους σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. So, just, just as a transition into innovative financial instrument, uh, Για αυτό το λοιπόν το καινοτόμο ε, πιστοτικό εργαλείο ήθελα να δω πώς συνδέονται οι επιδοτήσεις που υπάρχουν μέσω αυτού του μηχανισμού και πώς θα συνδυαστούν με έργα κοινού ενδιαφέροντος όπου θα δώσουμε την ε, προστιθέμενη αξία την ευρωπαϊκή. Γιατί θα πρέπει να δούμε αν το ιδιωτικό κεφάλαιο μπορεί να μοχλευθεί πριν να προχωρήσουμε σε διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και νομίζω ότι αυτά τα καινοτόμα μέσα είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα και χαίρομαι που βρίσκονται στον πυρήνα του ίδιου σας του έργου. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πριν ε, θεωρήσετε πως αυτά τα καινοτόμα ε, επενδυτικά μέσα είναι αποτέλεσμα μαύρης μαγείας, όπως είπε ο συνάδελφος, να σας εξασφαλίσω πως αυτά τα εργαλεία τα χρησιμοποιούμε από τη δεκαετία του 90. Ε, κυρίως ως εγγυήσει ε, είτε για κεφάλαιο κινδύνου είτε για μικρομεσές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ακολουθούμε κάποιες πολύ δοκιμασμένες ε, επενδυτικές τεχνικές και το καινοτόμο δεν είναι ότι προτείνουμε τη χρήση τους, αλλά πως προτείνουμε να επεκταθεί η δράση τους σε νέους κλάδους και με πιο συντονισμένο τρόπο. Δεν θα ήθελα λοιπόν να νομίζετε εδώ πως κάνουμε κάτι το ριζικά ανατρεπτικό. Όχι, θα οικοδομήσουμε αυτές τις προσπάθειες πάνω στη βάση των περασμένων επιταχειών. Αυτό λοιπόν, ε, το, αυτός ο μηχανισμός του CEF θα χρησιμοποιήσει εργαλεία τα οποία είχαμε από το παρελθόν το equity όπως επίσης και το μηχανισμό κατανομής ε, κινδύνου. Έχουμε γύρω στα δύο δις για τις μεταφορές, ένα δις για την ενέργεια και κάτι παραπάνω για την κοινωνία των πληροφοριών, ε, κονδύλια τα οποία έχουν ε, χρησιμεύσει στο παρελθόν και τα οποία μπορούν να επαναπροσανατολιστούν προς αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει κάποιο εταίρο όπως θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το EIF ή κάποιοι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ε, σύμφωνα με τα όσα θεσπίζει ο σχετικός ε, κανονισμός. Με τις προτάσεις όμως που καταθέτουμε εδώ είναι πρώτα απ' όλα η δημοσιονομική δέσμευση που κάνουμε ε, όπως κάνουμε για οποιαδήποτε άλλη επένδυση και αυτό θα πληρωθεί στον, ε, εφαρμοστικό, στον εταίρο που εφαρμόζει, που υλοποιεί το έργο. Άρα λοιπόν η δική μας συμβολή, συμβολή σε αυτό το πιστοτικό εργαλείο ε, έχει ως ε, την, το ποσό που έχει δεσμευτεί στον προϋπολογισμό από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το δεύτερο είναι πως αυτά τα εργαλεία, επειδή επιτρέπουν να προσελκυθούν και άλλα κονδύλια ε, στις επενδύσεις αυτές και από τις αγορές και από άλλους επενδυτές, ίσως και από τις τράπεζες, έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να αυξηθεί το τελικό ποσό ε, χρηματοδότησης προς τον τελικό ε, δικαιούχο. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάτε για πολλαπλασιαστικό παράγοντα ή για μόχλευση, δεν θα ήθελα να δαιμονοποιήσουμε, αλλά είναι μια μικρή συμβολή του ευρωπαϊκού προπολογισμού που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αυξημένα τελικά ωφέλη, επαναλαμβάνω για τον τελικό δικαιούχο. Και το βέβαια τελικό πλεονέκτημα είναι η ευελιξία που προσφέρει, γιατί στοχεύει, ε, είναι στοχευμένο ε, κεφάλαιο, ε, το οποίο έχει το σωστό μείγμα στις σωστές αναλογίες για το σωστό κεφαλαίο, για το σωστό σχέδιο. Η άλλη διαφάνεια αναφέρεται στις αρμοδιότητες. Δεν θα σχολιάσω σε βάθος. Νομίζω ότι η οικονομική εφαρμογή ε, επαφίεται στον ανάδοχο και αυτό βέβαια θα γίνει όταν τα χρηματοπιστωτικά αυτά μέσα βρεθούν στη βάση της ορίμανσης. Οπότε και οι τράπεζες ή ο χρηματοδοτικός εταίρος θα αποφασίσει κατά πόσο το σχέδιο το οποίο υποβάλλεται προσέγγιση ε, θα ενταχθεί ή όχι. Αυτό επιτρέπει και μια διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και σε επίπεδο σχεδίων αλλά και σε επίπεδο γεωγραφικό. Και η τελευταία διαφάνεια που έχει να κάνει με τα ε, ε, εργαλεία αυτά, που είναι τα ομόλογα έργου, είναι το εργαλείο το οποίο πιο πολύ έχει ε, προχωρήσει σε επίπεδο του Connecting Europe Facility, του CEF και μάλιστα έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ που προτείνουμε να περάσουμε και σε μια φάση πιλωτική για το 2012-2013 το προτείνουμε γιατί έχουμε συσσωρεύσει εμπειρία τα τελευταία χρόνια και με το σύστημα εγγυήσεων για τις ε, μεταφορές που συνεργαστήκαμε με τη σχετική Γενική Διεύθυνση και είδαμε πως χρειάζεται τελικά αρκετός χρόνος για τους διάφορους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντας σε ένα ε, έργο ε, να εντάξουν νέα εργαλεία στις χρηματοπιστωτικές τους αποφάσεις. Στο εργαλείο που έχουμε για τις μεταφορές έχουμε πάντα κάποιους χορηγούς έργων όπου όσοι χτίζουν γέφυρες, δρόμους, μέσα σταθερές τροχιάς, ποθήκες δεξαμενές αερίου, χρηματοδοτούνται από τράπεζες. Με αυτά τα ομόλογα έργου θα ακολουθήσουμε την ίδια τεχνική χρηματοδότησης και θα την επεκτείνουμε και δεν θα έχουμε μόνο τραπεζικά δάνεια, αλλά θα έχουμε και έκδοση ομολόγων ε, χρηματοδότησης συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Τι σημαίνει αυτό. Έχουμε, ανοίγει η γκάμα των εταίρων που έχουμε, δηλαδή επενδυτές, για παράδειγμα ασφαλιστικά ταμεία, ταξιδοτικά ταμεία, έτσι ώστε όλοι αυτοί να εξοικειωθούν με το προϊόν μας. Ε, και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε την πιλωτική φάση, αντί να περάσουμε τα πρώτα δύο χρόνια ε, της ε, φάσης εφαρμογής, τελικά για να αποκτήσουμε το ίδιο πλεονέκτημα. Την εξοικείωση δηλαδή με το εργαλείο αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε την πιλωτική φάση με ήδη υπάρχοντα κονδύλια Έχουμε τα 200 εκατομμύρια από, το, από τις μεταφορές, 10 από την ενέργεια και 20 από την κοινωνία της πληροφορίας και με αυτά τα ποσά θα προχωρήσουμε. Βέβαια είναι περιορισμένα τα ποσά, περιορισμένος ο χρόνος, όσο και να προσπαθήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την πιλωτική φάση δεν θα πάμε πολύ γρήγορα και θα έχουμε μόνο ε, μερικά έργα που θα προχωρήσουν έτσι. Παρ' όλα αυτά θα δώσουν πολύτιμη εμπειρία και επαναλαμβάνω θα μας εξοικειώσουν όλους με αυτή τη νέα έννοια που είναι τα ομόλογα έργου και το πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στην πράξη. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όντως υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση την οποία ανέφερα εν συντομία προηγουμένως και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να τη συζητήσουμε και με βάση τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα όμως, ολοκληρώνοντας, να πω ότι όσον αφορά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, παράδοξα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά χρήματα στην αγορά σήμερα για τέτοιου είδους έργα. Και η πρόκληση ποια είναι για αυτούς που προωθούν το έργο αυτό, είναι να μπορέσουν να συγκεντρώσουν, να χαλιναγωγήσουν αν θέλετε όλα αυτά τα χρήματα για να, μπορέσουν, ε, να μπορέσουμε να έχουμε project υψηλότερης ποιότητας και υψηλότερης ε, προστιθέμενης κοινωτικής αξίας. Πιστεύουμε ότι αυτό το εργαλείο θα μπορέσει να ε, τραβήξει τα κεφάλαια αυτά. Θα, από πλευράς της Κομισιόν θα είμαστε σίγουροι ότι με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές θα μπορέσουμε να πείσουμε, αν θέλετε, και τους αυτούς που προωθούν το έργο, τους υπεύθυνους του έργου, να ε, σεβαστούν όλα τα κριτήρια. Και θέλουμε, ούτως ή άλλως, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, να έχουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο επειδή όμως υπάρχει και μια δημοσιονομική, δημοσιονομική πειθαρχία, θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές όσον αφορά τα project. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι η δομή των project είναι απόλυτα εστιασμένη και ότι μπορούν να εφαρμοστούν και να χρηματοδοτηθούν κάτω και από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολλές πληροφορίες λάβαμε, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ήδη έχουμε και έναν μακρύ κατάλογο ομιλητών και μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό που θα δημιουργηθεί γιατί είναι πολλές ερωτήσεις και είναι και πολύ διαφορετικά τα θέματα. Λοιπόν, για να δω δύο λεπτά ποιοι έχουν δηλώσει. Για να... Ε, λοιπόν, να... μια που δεν έχουμε εισηγητή, Όποιος πήρε, όποιος ε, σήκωσε πρώτο στο χέρι του θα πάρει και, την, και πρώτο τον ε, λόγο. Ο κύριος Σιωμάνσκι έχει όπως πάντα ζητήσει πρώτο τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Διάβασα την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για το CEF, το Connecting Europe Facility. Άκουσα και τις παρουσιάσεις των προσυκλημένων και είναι σαφές ότι όλες οι ε, επενδύσεις για την ενέργεια θα βασιστούν σε δύο πράγματα. Επενδύσεις σε, νέες, ε, σε νέους διαδρόμους ενέργειας, κυρίως για την κεντρική Ευρώπη, που θα επιτρέψουν και τον ανταγωνισμό στον τομέα της, ε, στην αγορά του αερίου και από την άλλη επενδύσεις που θα γίνουν για την για να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους ας πούμε, η σύνδεση των αιωλικών πάρκων στον νότο και των φωτοβολταϊκών πάρκων στο βορρά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η Κομισιόν έχει κάνει κάποια μελέτη που να δείχνει έτσι μια αναλογία μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων τομέων επενδύσεων. Δηλαδή, μπορείτε να μας, δει, να μας δώσετε κάποια χοντρικά νούμερα για το ποια θα είναι τα ποσά που θα δαπανηθούν σε αυτούς τους δύο τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους και τις εκπροσώπους από την Κομισιόν. Ήταν πολύ χρήσιμες οι παρουσιάσεις τους, έτσι για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το πώς έχει η κατάσταση. Πρώτη παρατήρηση. Τα, τα οράματα χωρίς να έχουμε επενδύσεις είναι μόνο ψευδεστήσεις τελικά και νομίζω ότι το CEF είναι μια πολύ καλή συγκεκριμένη πρόταση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ευρωπαϊκά μεγάλα project στην Ευρώπη και να έχουμε και, μια που δεν έχουμε ενιαία αγορά, να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτού του ε, στόχου. Βασικά λοιπόν θεωρώ ότι η πρόταση είναι πολύ θετική. Δεύτερον, δεν, είναι, δεν μου είναι απόλυτα σαφές τι θα γίνει με αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν ξέρω πώς, πόσο το, σίγουρο είναι η Κομισιόν γι' αυτό. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διάφορες συζητήσει για διάφορα οικονομικά πλαίσια, για διάφορα πολυ, πολυετή προγράμματα, για το ενέρευνα, για, την, για, το γεωργικό, για τον προπολογισμό για τη γεωργία. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδυαστούν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα 50 δις, για να είναι λίγο σαφές το πράγμα, για μένα τουλάχιστον, είναι το σύνολο των επενδύσεων που θα γίνει από ανακατονομή ας πούμε άλλων γραμμών α, του προπολογισμού συν δάνεια, συν ομόλογα ε, αυτό είναι το ποσό αυτό το 50 δις γιατί μιλήσατε για 50 δις που θα πάνε στους τρεις αυτούς τομείς. Είναι το συνολικό ποσό που θα υπάρξει για επενδύσεις ή εγώ δεν κατάλαβα πολύ καλά και πρέπει να ξεπεράσουμε και το ποσό αυτό. Μετά, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μπορούμε να πούμε πολλά και θα ήθελα να δω αν υπάρχουν αξιολογήσεις στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ήδη χρησιμοποιούμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Το risk and sharing, τα, ε, η ε, συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων, ειδικά όταν μιλούμε και για την τράπεζα επενδύσεων. Υπάρχουν κάποιες αξιολογήσεις, κάποιες αξιολογητικές εκθέσεις από τις οποίες να έχετε καινούργια συμπεράσματα για τα ομόλογα τώρα. Ε, ποιος, έχει την ε, ηγετική θέση ας πούμε, ποιος είναι ο οδηγός. Αυτά τα ομόλογα είναι, των έργων είναι ομόλογα που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα, η, η Κομισιόν έχει τον ηγετικό ρόλο, αυτή το διαχειρίζεται, αυτή το ελέγχει ε, με όλη τη διαδικασία ας πούμε, της καλής διακυβέρνησης ή έχει τη διακυβέρνηση της, του project. Τι ακριβώς γίνεται, αν μπορούσατε να μας πείτε δύο πράγματα και γι' αυτό θα με βοηθούσατε πολύ. Μετά, για το ICT. Ε, ζητώ συγγνώμη που έχω τόσες πολλές ερωτήσεις, αλλά κλείνω. Ε, η συνάδελφό σας είπε ότι με, το, με τη σωστή προσέγγιση στην, στον κανονισμό, σε μια ρύθμιση, μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Μήπω μπορείτε να το κάνετε αυτό λίγο πιο σαφές. Πού υπάρχει το πρόβλημα τελικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τι θα πρέπει να βελτιωθεί. Πού βρίσκονται τα προβλήματα, τα διέξοδα τα οποία έχουμε και ώστε να μπορέσουμε να, το, να έχουμε διευρυζωνικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη θα κλείσω για να, πούνε και άλλοι, να πάρουν και άλλοι το λόγο, αλλά η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, έχει εμπλακεί καθόλου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν ε, και στα κράτη-μέλη, ε, υπάρχει προς τα κράτη-μέλη χρηματοδότηση για την επίτευξη αυτών των, αυτών των προγραμμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει εμπλακεί και αν υπάρχει σύνδεση και με, τις, με την Γενική Διεύθυνση αυτή γιατί υπάρχει και μια πρώτη διαδικασία clearing ε, και μια διαδικασία μετά κοινοποίηση που πρέπει να υπάρξει. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν κάποιε διευκολύνσει ή πώ ακριβώ ε, έχετε συνεννοηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Σαουντάκα. Ε... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για, την, ε, για τις παρουσιάσεις σας γιατί εγώ προέρχομαι από μια χώρα της Βαλτικής, από την Λιθουανία και εκτιμώ ιδιαίτερα την Κομισιό και τον Επίτροπο στην, στον τομέα ενέργειας διότι όντως το το θέμα της ενέργειας είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες επί, ε, μας. Επειδή όμως πρέπει να φύγω γιατί σε μια άλλη επιτροπή πρέπει να ψηφίσω, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ε, την αποκοπή που πρέπει, θα πρέπει κάπως να αποσυνδεθούμε σαν χώρες της Βαλτικής από την Ρωσία διότι έχουμε ε, άμεση ας πούμε, σύνδεση με, το, με τα ηλεκτρικά δίκτυα με την Φιλανδία, με τη Σουηδία, με την Πολωνία και αυτά τα project πρέπει να προχωρήσουμε. Γίνονται όμως και μελέτες κοπιμότητες οι οποίες ε, θα ολοκληρωθούν ε, την ε, επόμενη χρονιά όπου θα υπάρξει ο αποσυγχρονισμός αν θέλετε από την Ρωσία και ο συγχρονισμός μας σαν χώρες Βαλτικής με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα αναφέρονται ρητά σε αυτό το, το CEF διότι χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο γιατί υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους γειτονές μας Ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία project για ολοκλήρωση τριών πυρηνικών ε, κέντρων ε, στην Λευκορωσία, στην Λιθουανία και στο Καλίνιγκραντ συνεργασία των τριών ε, αυτών χωρών. Και αφού αποσυγχρονιστούμε από την Ρωσία θα δημιουργήσουμε έναν άλλο νησί αν θέλετε για την Ρωσία διότι η περιοχή του Καλίνιγκραντ θα είναι ένα νησί όσον αφορά το συγχρονισμό. Αυτά όμως τα θέματα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και ζητώ συγγνώμη που αναφέρθηκα σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για μας είναι ζωτική σημασία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι ήρθε στη συνεδρίασή μας και μάλιστα με τόσους πολλούς εκπροσώπους για να μας πει με τέτοια σαφήνεια ε, ποιε είναι οι προθέσεις της. Και μάλιστα ήταν και εξαιρετικά σαφές και το κείμενο το οποίο κατέθεσε. Είναι ένα κείμενο και ένα πακέτο προτάσεων πολύ σημαντικό. Βεβαίως και έχουμε το χρόνο, το συζητήσουμε σε βάθος από εδώ και στο εξή και σήμερα θα ήθελα μετά από μια πρώτη γρήγορη ανάγνωση να αναφερθώ σε ένα από αυτά τα ε, σημεία, τα οποία βέβαια εσείς ξεκαθαρίσατε στις παρεμβάσεις γιατί στο κείμενο δεν το είχα καταλάβει. Πιο συγκεκριμένα είναι το πρώτο παράρτημα ε, στο, σχετικά με την ενέργεια έγγραφο, γιατί διαβάζοντάς το ε, αισθάνθηκα μεγάλη έκπληξη και μετά βέβαια από τα λεγόμενά σας ακόμα περισσότερο, διαβάσοντας πως η Ιβηρική Χερσόνησος, γιατί το είπατε και εσείς, είναι ένα πραγματικό, ε, μια πραγματική νησίδα εκτός ε, ευρωπαϊκών δικτύων ε, και αναφέρεται μαζί με άλλα κράτη-μέλη στο εδάφιο που αναφέρεται στην διασύνδεση βορρά-νότου με κοινό στόχο να έρθει ανανεώσιμη ενέργεια από την Αφρική στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό αυτό. Μήπως όμως θα έπρεπε να αναφερόμαστε και ρητά στις χώρες αυτές, μια και επίγει το θέμα σήμερα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως η διασύνδεση της Ιβηρικής Χερσονήσου θα ξεκινήσει από τη διασύνδεση με τη Γαλλία, γιατί αυτό λείπει από το κείμενο και για το φυσικό αέριο. Ε, δημιουργήθηκε και μία σύγχυση όταν το διαβάζαμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ένα στιάδρομο φυσικού αερίου από τον νότο ή ε, από τη Δύση ε, θα ε, μπορούσε να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό μέσω των Πυρηναίων με πολύ πιο φθηνό τρόπο από όταν επιλέξουμε κάποιες άλλες διαδρομές. Αυτό μας λένε άλλωστε και οι σύμβουλοι μας που ξέρουν τα θέματα της αγοράς. Γιατί λοιπόν ε, αυτό δεν φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στο πρώτο παράρτημα. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημά μου, αλλά επειδή επηρεάζει άμεσα τη θέση της χώρας μου, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες συγκεκριμένες εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Μια που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα, θα έλεγα να κάνουμε ένα, μια παύση εδώ, γιατί ήταν πολλέ οι ερωτήσει και είναι και διαφορετικοί οι τομεί. Να δώσουμε την ευκαιρία στου ε, προσκεκλημένου μα να απαντήσουν. Ε, νομίζω ότι επειδή είναι τόσε πολλέ οι ε, ερωτήσει, μετά θα μπερδευτούμε τελείω. Οπότε για να έχετε και εσεί τι αφήσει σα απαντήσει, σα δώσουμε πρώτα το λόγο στου καλεσμένου μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ χρήσιμο το διάλειμμα που κάνετε. Να σας ενημερώσω λίγο για την εμόχλευση και για τα 50 αυτά ό,τι αφορά τι επενδύσεις. Ε, είναι διαφορετικό βέβαια σε αυτό ανάλογα με τον τομέα και στην ενέργεια και στα ψηφιακά θέματα θα ακούσετε τα αριθμητικά στοιχεία από τους συναδέλφους. Ε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να κάνουμε έτσι μια πλήρη εκτίμηση γιατί θα εκτιμηθεί από το πώς θα προετοιμαστούν τα προγράμματα, τα έργα, πώς θα παρουσιαστούν και ποιο θα επιλεγεί τελικά. Αλλά η βασική προετοιμασία για, τα, για τις επιδοτήσεις αυτές και για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχει ως στόχο να ενισχύσει τη μόχλευση. Ας πούμε, για, τον, για τις μεταφορές, τον τομέα των μεταφορών και το παράρτημα που αφορά τις μεταφορές, όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός projects, η συνολική επένδυση που σχετίζεται με αυτά τα project είναι περίπου 220-230 δις για, το, για τις μεταφορές. Και θεωρώ ότι με το 31,7 μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό τον κατάλογο των projects. Κάποια projects προφανώς δεν θα έρθουν, κάποια θα είναι μικρά, κάποια θα είναι μεγαλύτερα, αλλά στο τέλος ο, το μέγεθος αυτών των, αυτών των επενδύσεων είναι επαρκές. Το 31,7 δηλαδή μπορεί να καλύψει τα έργα αυτά θα εξαρτηθεί βεβαίω και, από και από την ποιότητα των projects, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να έχουμε δηλαδή έναν κατάλογο που να είναι συμμορφούμενο με, ε, με το παράρτημα. Οπότε εκεί, αυτό είναι, αυτή η μόχλευση προβλέπεται για του τομεί αυτού και για, τα, για, τα, για την επιδότηση, αλλά και για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ε, να μα πείτε εσεί για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μετά οι συνάδελφοι. Mm the 230 as well. No, just the evaluation and uh, the project bonds within the mm. driving seat. Um, um, well, uh, κοιτάξτε. Για την αξιολόγηση των υπαρχών των δημοσιονομικών εργαλείων. Δύο από τις αξιολογήσεις, μία του SSF και, και το EIB, όλη η αξιολόγηση των ε, για τα δάνεια, για τα για εγγύησεις ε, που δίνει το, για τα ΤΕΝ έχει ολοκληρωθεί. Φαίνεται ότι κάπου βέβαια οι αξιολογήσεις αυτές ε, σε ηλεκτρονικό επίπεδο έχουν χαθεί, θα το βρούμε, θα τις βρούμε όμως και θα γίνει μια βέβαια περαιτέρω ολοκληρωμένη μελέτη του LGTT, αλλά για, τα, για την πρωτοβουλία των ονομολόγων έργου, που είναι, αν θέλετε, η, η ναυαρχίδα μας, ας πούμε, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Κομισιόν βέβαια. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα οποία θα πληρωθούν ε, στον, στον Ευρωπαίο, αν θέλετε, υπεύθυνο του project και αυτό μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από εκεί θα πληρωθούν τα ομόλογα. Δηλαδή είναι μακριά η αλυσίδα, αλλά αυτός ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο είναι αυτός ο οποίος θα εκδώσει τα ομόλογα. Και το έργο του δημοσιονομικού εταίρου ή της Κομισιόν ή της Τράπεζας είναι να διευκολύνει την όλη διαδικασία να ολοκληρώσω αυτό, γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό πώς ε, χρησιμοποιείται η κοινοτική χρηματοδότηση και πώς θα γίνει η χρηματοδότηση των project με πιο ε, εύκολο τρόπο. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία έχουν μια κάποια προϊστορία και το LGTT και στις μεταφορές η Κομισιό έχει αποκτήσει κάποια εμπειρία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μέσω της δημιουργίας ενός ε, κέντρου εμπειρογνωμοσύνης ε, του EPP και ε, στις περιοχές μας έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τους, αυτούς που προωθούν τα έργα, τα διάφορα project. Δεν χρηματοδοτούνται όλα αυτά με μαγικό τρόπο τρόπο, το ξέρουμε. Είμαστε όμως σίγουροι σχεδόν ότι μπορούν να προωθηθούν αν θέλετε τα project αυτά, διότι την ευθύνη την έχει αν θέλετε τόσο ο οποίος προωθεί το project και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και η πρόκληση για την Κομισιό είναι να εξασφαλίσει ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των project έχουν στρατηγική σημασία για την ολοκλήρωση την, της ημερήσιας διάταξης, αν θέλετε, και των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στους τρεις αυτούς τομείς. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις όσον αφορά την ενέργεια. Θα ξεκινήσω με τις, με τις ανάγκες τις επενδυτικές και για τα ποσά. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο έχουμε υπολογίσει ότι θα πρέπει να επενδυθεί από σήμερα μέχρι το 2020, αλλά εδώ μιλάμε για παραγωγή, για κατανομή, όλο το, το φάσμα αν θέλετε των επενδύσεων. Αυτό το οποίο εξετάζουμε εδώ στην πρότασή μας ε, είναι ποιες ε, είναι οι ανάγκες ε, για τις επενδύσεις στην στις, ε, στη μεταφορά του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 200 δισεκατομμύρια μέχρι το, 2000, ε, ε, μέχρι το 2020 140 για τον, για, την, για τον ηλεκτρισμό και 70 περίπου για, την, για το αέριο. Από αυτά τα 200 δισεκατομμύρια, με, σύμφωνα με, τον, με το υπάρχον ε, σύστημα ε, κανονιστικό, το κανονιστικό πλαίσιο, θα έχουμε μία εφαρμογή χωρίς προβλήματα, business as usual, και μετά τα 50 δισεκατομμύρια θα καθοστορήσουν εξού και η πρότασή μας να υπάρχει μια επιτάχυνση μέσω των επιχορογήσεων. Επομένως το CEF ε, δίνει 50 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις που δεν πρόκειται να ε, υλοποιηθούν λόγω δυσκολιών πρόσβασης ή γιατί το 1,1 δισεκατομμύρια της ενέργειας που δίδεται στην ενέργεια έχει υπολογιστεί με βάση την, την μόχλευση μέσω των ε, επιχορηγήσεων ή μέσω δημοσιονομικών εργαλείων έτσι ώστε να καλύψουμε το κενό των 50 δισεκατομμυρίων που, μπορεί, που θα δημιουργηθεί και, και το οποίο δεν θα δημιουργεί το αν υπήρχε δημόσια δράση. Ο, δεν τίθεται ούτω ή άλλω και θέμα ανταγωνισμού λόγω τη συνεργασία ανάμεσα στον ειδικό και στον δημόσιο τομέα. Τώρα, όσον αφορά την, τον αποσυγχρονισμό των ε, χωρών της Βαλτικής από το ρωσικό σύστημα η Κομισιόν θα προτείνει μια διαπραγματευτική εντολή σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ε, διαδικασία αυτή, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και τεχνική χαρακτήρα. Ε, δεν μπορεί να φύγουμε άμεσα και απότομα από το ρωσικό σύστημα διότι θα έχουμε ένα blackout στις χώρες της Βαλτικής αλλά ε, συνεργαζόμαστε με το ευρωπαϊκό σύστημα των ε, επιχειρήσεων στον τομέα του, του ηλεκτρισμού έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνδέσεις ανάμεσα στις χώρες της Βαλτικής και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουμε και συζητάμε με τους Ρώσους τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι συνδέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ρωσία αλλά και ανάμεσα στις χώρες Βαρτικής και στο Καλίνιγκραντ. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία διότι ο ηλεκτρισμός είναι περίπλοκο πράγμα. Τώρα, όσον αφορά αυτή την εισίδα, την ενεργειακή στην οποία αναφερθήκατε και που είναι η Βυρική Χερσόνησος. Για μας η, η Βυρική Χερσόνησος θα έπρεπε να το ξεπεράσει και δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη σύνδεση και για το φυσικό αέριο και για τον, ε, την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι μια προτεραιότητα για το 2014-2015 και νομίζω πως αυτό θα επιτρέψει και στην Ευρώπη ε, μετά τη Γαλλία, προς, ε, εννοώ και στις χώρες ε, πιο βόρεια από τη Γαλλία, να χρησιμοποιήσουν το όφελος και το πλεονέκτημα που προσφέρει η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας στην Ισπανία. Γι' αυτό έχουμε προτείνει και μια περιφέρεια η οποία επεκτείνεται και πέραν της Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και κάποια κράτη-μέλη που είναι πιο βόρεια μια και εκεί θα πρέπει να γίνει η διάθεση ε, και η αντιστοίχηση ε, του ε, της παραγωγής από ΑΠΕ με την ζήτηση για ενέργεια από ΑΠΕ για τις χώρες της Βορειοαφρικής μιλάμε για μια πιο μακροπρόθεσμη ε, προτεραιότητα η οποία προσεγγίζει τον ορίζοντα του 2020. Σας εξασφαλίζω όμως και σας εγγυώμαι πως για μας προτεραιότητα είναι η διασύνδεση της Ιβυρικής Χερσονήσου το συντομότερο ε, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα στην περίοδο του 2014-2015. Για να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε ε, για τον ε, κλάδο των τηλεπικοινωνιών, να σας πω πως δεν ξέρω να έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να τοποθετηθεί κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο διαφορετικό από αυτό το οποίο ισχύει από τη δεκαετία του 90 και αναθεωρήθηκε πριν από δυόμιση χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα και το κόστος της τηλεφωνικής κλήσης στην Ευρώπη έχει πέσει τουλάχιστον 40% από την απελευθέρωση των αγορών. Αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι πως οι επενδυτικές δραστηριότητες των ε, εταιριών τηλεφωνίας ε, έχει επιβραδυνθεί. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια άρθρα από το ρυθμιστικό πλαίσιο γιατί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού δεν είναι βέβαια αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ανεξάρτητες οι ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές μέσω του συντονιστικού έργου που είναι το Μπάρακ και βέβαια εκδίδουμε συστάσεις. Όταν λοιπόν μίλησα για μια αύξηση της ρυθμιστικής ασφάλειας και βεβαιότητας έτσι ώστε να είναι πιο καλό το επενδυτικό κλίμα αναφερόμουν στις προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή για την, για την μεθοδολογία κοστολόγησης και για την απρόσκοπτη πρόσβαση που αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση. Εδώ δεν μπορώ να σας δώσω κάποιες απαντήσεις για την ε, βελτίωση αυτών των κειμένων. Χρειαζόμαστε βέβαια κάποιες, ε, κάποιες προσανατολιστικές οδηγίες για το πώς μπορούν να βελτιώσουν το όφελος και για τον καταναλωτή ρυθμιστικές αρχές, αλλά και για τους επενδυτές που πρέπει να καλύψουν και το κόστος της επένδυσης, αλλά και τον κίνδυνο που ενέχει κάθε επένδυση. Εμείς, ε, επαναλαμβάνω, επεμβαίνουμε μέσω μιας ε, προσέγγισης η οποία επιτρέπει να υπάρχουν επαρκή κεφάλαια επενδυτικά, το οποίο τι σημαίνει επαρκή σε ύψους, αλλά τα οποία αναγνωρίζουν και την ανάγκη ορίμανσης των επενδυτικών σχεδίων, όπως και τις πολυπλοκότητες χρηματοδότησης αυτών. Δηλαδή, η ορίμανση φέρνει ε, του, την επιτυχία και είναι ένα θέμα το οποίο ε, παρακολουθούμε παράλληλα με τις υπόλοιπες πτυχές του εργαλείου μας. Τώρα για τις κρατικές επιχορηγήσεις, κρατικές επιδοτήσεις και τον ανταγωνισμό, η αγορά απελευθερώθηκε στις τηλεπικοινωνίες ε, και στην χρήση και στις υποδομές αλλά ακόμα αρκετοί παίκτες έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς όπως επίσης έχουν και πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη από την εγκατάσταση των δικτύων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη που όμως δεν προσφέρουν άμεσες ε, οικονομικές αποδόσεις. Άρα λοιπόν οι δημόσιες αρχές έχουν συμφέρον να εξασφαλίσουν πως τα δίκτυα αυτά υπάρχουν παντού. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση για τη δημιουργία, ε, για την εγκατάσταση μάλλον επιχειρήσεων σε μια περιοχή. Αν ρωτήσει κανείς, και συνεχώς ρωτάμε τις επιχειρήσεις, για ποιο λόγο θα πηγαίνατε κάπου, μας είπαν αυτό το οποίο θα μας οδηγούσε σε μια μετεγκατάσταση ενδεχομένω είναι ε, η υψηλής ταχύτητας ε, διασυνδέσεις. Επτά από, τις, από τα ΣΔΙΤ που αναλύσαμε, όπου το δημόσιο ε, προσφέρει τα κονδύλια έτσι ώστε να εγκατασταθούν αυτά τα υψηλής ταχύτητας δίκτυα, ε, γίνεται μέσω κρατικών, επιχειρη... Ε, γίνεται μέσω κρατικών επιδοτήσεων. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, οπωσδήποτε περνάνε από τη διαδικασία έγκρισης κρατικής επιδότησης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Όμως, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές επιδοτήσεις που έχουν ε, διατυπωθεί ακριβώς για το θέμα της ευρυζωνικότητας, είπαμε χρειάζεται συνέχεια και της δημόσιας στήριξης των δημοσίων υποδομών και όλων των υποδομών, γιατί βέβαια το πιο ακριβό τμήμα της επένδυσης είναι, πιστέψτε, οι εξκαφές και θα πρέπει εδώ οι εξκαφές αυτές να γίνονται παράλληλα έτσι ώστε να εγκατασταθούν όλα τα δίκτυα υποδομών. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση για όλων των εταιριών στους αγωγούς ε, γιατί πολλές φορές οι διάφορες επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές τους από την ε, δυνατότητα αυτή μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι βεβαίω ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ ώστε να υπάρξουν στο δυνατόν περισσότερα κονδύλια. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολλά δημόσια κονδύλια. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα πολλαπλασιάσουμε τα λεφτά που έχουμε. Αυτό είναι κατανοητό. Βεβαίω και τα εργαλεία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν. Και θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω, είπατε ότι κάποια από αυτά τα εργαλεία ήδη υπάρχουν. Είπατε ότι δίνονται στους εταίρους μας χρήματα και τα χρησιμοποιούν. Δεν υπήρξαν ε, ερωτήματα για το αν υπήρχε επαρκής έλεγχος στο παρελθόν. Δηλαδή, έχει γίνει χρηστή διαχείριση ας πούμε, αυτών των κονδυλίων. Δεν το έλεγξε ποτέ κανείς αυτό. Ε, θα ήθελα μια απάντηση. Μπορεί να είναι μια δική μου χαζή ανάμνηση βέβαια. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ σημαντική συζήτηση για το πώς γίνεται ο έλεγχος των κονδύλιων αυτών από την Κομισιόν. Ε, μπορεί να υπήρξαν κάποια προβλήματα, ναι. Αλλά η μονάδα για την, για την έρευνα έκανε μία μελέτη ακριβώς για τη συγχρηματοδότηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ο έλεγχος, ότι όλα έγιναν ε, τελικά σωστά. Ωραία. Να αφήσουμε λοιπόν και τους υπόλοιπους συναδέλφους να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι αντιμετώπισα με μεικτά αισθήματα την ανακοίνωση αυτή διότι ανήκω σε μια ομάδα βουλευτών που βρισκόμαστε στην ε, μειοψηφία όταν παρουσιάστηκαν οι στόχοι του 2020. Διότι είπαμε μπει και στον πρόεδρο Μπαρόζο ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο σχέδιο επενδύσεων. Και όταν είδαμε την ανακοίνωση της Κομισιόν, είπαμε να, εδώ έχουμε ένα μεγάλο project που μέσα στα πλαίσια ε, των ε, προσπαθειών ε, των κυβερνήσεων να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, μια και αρχίζουμε και διώχνουμε τα λιγότερα, τις λιγότερο αξιόπιστες κυβερνήσεις, ε, προσπαθούμε να πετύχουμε την ε, ανάπτυξη την οποία να έχουμε ανάγκη. Και πώς θα γίνει αυτό, προωθώντας την εσωτερική αγορά, την, την απασχόληση και όλα αυτά με ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών. Αυτό το κάνουν. Όλοι το κάνουν σε όλο, το, το, την, σε τον πλανήτη. Η Βραζιλία το κάνει. Έχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία. Και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα σύνδεσης στην Ευρώπη. 50 δισεκατομμύρια. Τι να σας πω. Πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν είναι στο ύψος ε, των περιστάσεων. Και το λέω έτσι όπως το αισθάνομαι, διότι σας ε, ε, βλέπουμε να διστάζετε όσον αφορά τις μεθόδους χρηματοδότησης. Είπατε ότι έχουμε στο παρελθόν εμπειρίες που λειτουργούν, θα δούμε. Και αναφέρω, αναφέρεστε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παντού. Μην τη χρησιμοποιείτε σαν συστατικό για όλες τις άλτσες. Πρέπει να έχει το, η τράπεζα αυτή έναν ε, εργαλείο, να είναι αποτελεί ένα εργαλείο συντονισμού. Μη δεν πρέπει να χάσει όμως πάση θυσία το, τα, τα τρία αλφα που έχει. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ δεν θα πρέπει να κάνετε προσπάθειες υπεργολαβίας και να διαχέεται η χρηματοδότηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι έχει την δυνατότητα να επενδύσει, διότι αν δεν αποδείξουμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε, ο ιδιωτικός τομέας δεν πρόκειται να επενδύσει. Ο ιδιωτικός τομέας επενδύει μόνο εφόσον επενδύει ο ε, δημόσιος τομέας. Μιλάτε για την πληροφορική, για την ενέργεια, για τις μεταφορές Υπάρχουν και άλλοι τρει τομείς όμως ε, που χρειάζεται επένδυση. Η... Το νερό, η πρόσβαση στο νερό θα είναι μια απέτηση των πολιτών μας και λυπούμε γιατί η, τροφοδότηση με νερό της Βαρκελώνας, ε, της Βαρκελώνας ε, μέσω μιας άντληση από τον Οροδανό έχει, είναι σε, σε στάση αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται υποδομές έρευνας και και το διάστημα. Αυτοί οι τρεις άλλοι τομεί. Και η ερώτησή μου είναι, η ερωτήση μου είναι Έχετε την πολιτική υποστήριξη των κρατών μελών, ε, γιατί τα κράτη-μέλη μας χρεοκοπούν αλλά παρόλα αυτά πολιτικά μπορούν να επηρεάσουν. Δεν είναι μόνο οι αλληλεσυνδέσεις. Εάν θέλουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων χρειάζεται και υποστήριξη ε, των κυβερνήσεων. τώρα, οι ρυθμιστές είπατε ότι δεν, χρειάζεται, δεν υπάρχουν χρήματα και όμως υπάρχουν χρήματα και εσείς το ίδιο το είπατε θα πρέπει στις καινοτόμες ε, χρηματοδοτήσεις ε, να βρούμε τις ε, σωστές εισφορές που δίνουν οι πολίτες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα σωστά project. Δηλαδή παίρνουμε από τον καταναλωτή και χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις. Αυτό το κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο, σε περιοχές όπου δεν μπορεί να παρέμβει, αν θέλετε, το, ο δημόσιος τομέας. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να ε, καθησυχάσουμε τους, πολί, τους πολίτες ότι εξυπηρετούνται από όλες αυτές τις προσπάθειες και ότι είναι ισότιμοι. Τώρα, οι κρατικές ε, ενισχύσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις ε, δεν χρειάζεται να τις συνεχίσουμε. Λέει η Κομισιόν Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χρηματοδότηση διότι είναι κρατική ενίσχυση. Αν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα είναι θα χάσει η, από την έγκλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτως ή άλλως ε, οι κρατικές ενισχύσεις μετά την Λισαβόνα είναι ένα μέσον αν θέλετε. Δεν είναι στόχος. Εάν χρειαζόμαστε κρατικές ενισχύσεις για να εξασφαλίσουμε την συνοχή του, του, της υπήρου μας, βρείτε έναν τρόπο να το εξασφαλίσετε. Μην κραδένετε αν θέλετε μπροστά στα μάτια των κυβερνήσεων τις κρατικές ενισχύσεις. Ζητώ συγγνώμη για το πάθος που δείχνω στην παρέμβασή μου, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβιβάσετε και σε όλους τους επιτροπούς και στον πρόεδρο της Επιτροπής ότι μέσα από αυτό το πρώτο βήμα, εδώ έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, κάποιος ποιητής είπε βέβαια ότι το πρώτο βήμα είναι και ένας ε, στόχος. Δεν ξέρω τέλος πάντων, αλλά τώρα αυτό το πρώτο βήμα που γίνεται, τώρα πρέπει να κάνουμε και τις επενδύσεις, ε, γιατί μετά από 20-30 χρόνια ε, θα είναι αργά πλέον για την ανταγωνιστικότητα του, της Υπήρου μας. Λοιπόν, με βάση αυτό το πρώτο βήμα θα πρέπει να μπορέσετε η Κομισιό, εσείς που κάνετε τις προτάσεις, αυτή είναι η δουλειά σας και η ευθύνη σας εξάλλου, θα πρέπει πρέπει να μας υποβάλλεται ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων. Ο συνάδελφος Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και περίκτικος. Ένα ερώτημα για την ε, διαδικασία διοδότησης, που είναι νομίζω από τα πιο σημαντικά στοιχεία και μάλλον από τα πιο αμφιλεγόμενα. Αναφερθήκατε σε ένα ανώτατο όριο τριών ετών για την ε, διοδότηση. Ε, οι άδειε αυτέ πρέπει να δοθούν από εθνικέ ή από περιφερειακέ, παύλα τοπικέ αρχέ των κρατών μελών. Ερώτημα. Πόσο υποχρεωτικό είναι αυτό, και υπάρχουν κάποια εργαλεία επιβολής κυρώσεων. Γιατί ας πούμε, αν μια εθνική αρμόδια αρχή που έχει ε, αναλάβει την εξουσία για να δώσει τις άδειες, δεν έχει δώσει την απαραίτητη άδεια στα πλαίσια αυτή της τριετίας, ας πούμε. Και όταν μιλούμε για ε, προγράμματα προτεραιότητας διασυνοριακά, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κύρωση σε αυτές τις εθνικές αρχές. Πώς μπορείτε δηλαδή να υποχρεώσετε να υπάρξει αδειοδότηση μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Γκίρεκ. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν διάβασα καλά το όνομά σα. Συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικές οι παρουσιάσεις που ακούσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε προστιθέμενη αξία στην, ε, στην κοινωνία των πληροφοριών, στην, ε, ε, στις μεταφορές και, στις, και στην ενέργεια. Πρέπει όντω να υπάρξει προστιθέμενη αξία και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Βεβαίω, ε, γι' αυτό χρειάζονται δάνεια ε, και χρειάζονται και σαφή κριτήρια για το πώ θα δοθούν κονδύλια στα ανάλογα, ε, στα ανάλογα προγράμματα. Και επίση, για ένα ερώτημα έχω να θέσω για τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα τη υπήρου μα. Κυρίω θα ήθελα να μιλήσω για, την, για τι μεταφορέ και κυρίω για την σύνδεση μεταξύ των, των κέντρων επιμελητίας και των μεταφορών. Γιατί η, αυτά τα, όσο πιο διεθνή είναι αυτά τα κέντρα, τόσο πιο ανταγωνιστική μπορούμε να γίνουμε κι εμείς. Και κυρίως εδώ μιλώ για κέντρα επιμελητίας τα οποία ας πούμε μπορούν να υπάρξουν στην Πολωνία ως διεθνή κέντρα. ή ας πούμε για να διευκολύνουν την, τις μεταφορές στην Ανατολική Ευρώπη. Ξέρουμε ότι τα κονδύλια για τις μεταφορές ε, μειώνονται και νομίζω ότι αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο παρόλα αυτά μπορούμε να έχουμε πολύ προστιθέμενη αξία. Και τώρα ο συνάδελφος Γκιούρεκ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν που και γραπτός και προφορικός μας έκανε τις παρουσιάσεις της. Όντως ε, είναι σωστές οι προτεραιότητες που προτείνονται ε, και τα εργαλεία. Ε, έχουμε όντως όμως πολλά προβλήματα στις αγορές αυτές, κυρίως όταν μιλούμε για την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Από την άλλη, Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση είναι το σημείο κλειδί και γι' αυτό δεν θα πρέπει εδώ τελευταία στιγμή ας πούμε, ή στην τελευταία μια μισή ώρα που μας έχει μείνει ε, να το αμελήσουμε το θέμα αυτό. Εγώ ε, ε, ενδιαφέρομαι πολύ για το θέμα της ε, ε, χρηματοδότησης, ειδικά όταν ε, μιλούμε για τον παράγοντα πολλαπλασιασμού και τις συνέπειες και το επίπεδο μόχλευσης που μπορούμε να έχουμε γιατί ξέρουμε ότι έχει υπάρξει μείωση των κονδυλίων της χρηματοδότησης και όλα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά. Αν τώρα όλο αυτό είναι λειτουργικό, είναι πρακτικό ή θα παραμείνει λειτουργικό και πρακτικό, μένει να το δούμε. Αλλά ε, η Κομισιόν φαντάζομαι πως ξέρει πού βρίσκονται τα προβλήματα και γι' αυτό και οι απαντήσεις που ακούσαμε μέχρι στιγμής ήταν σωστές και συνεκτικές. Ε, θα ήθελα να πω έτσι κάποια γενικά σχόλια για τη χρηματοδότηση ας πούμε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των, του Ταμείου Συνοχής και των υποδομών. Ξέρουμε ότι μιλούμε για 40 δισεκατομμύρια. Υπάρχει μια σχετική γραμμή του προπολογισμού που είναι διαθέσιμα, αλλά το ερώτημα είναι ε, υπάρχουν άλλα κονδύλια, μπορούμε να βρούμε άλλα κονδύλια για να συμπληρωθεί αυτό το ποσό. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα μπορούσα να σας θέσω. Ε, ο πρόεδρος βεβαίως μου πήρε και το, αυτό που ήθελα να πω από το στόμα και εγώ ήθελα το ίδιο ερώτημα να θέσω. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν χρηστά. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε. Και ένα τρίτο ερώτημα. η περιφερειακή διάσταση πώς λαμβάνεται υπόψη. Δεν μιλώ για την, για την ισορροπία μεταξύ της περιφερειακής και της εθνικής ή διασυνοριακής διάστασης, αλλά θα πρέπει και σε περιφερειακό επίπεδο να δούμε τι γίνεται, γιατί μιλούμε και για χώρες οι οποίες είναι πολύ φτωχές και η δυνατότητα χρηματοδότησης που έχουν είναι πολύ περιορισμένη. Οπότε θα ήταν καλό αυτές τις ανισορροπίες που υπάρχουν να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε υπόψη μας πολύ περισσότερο την α, περιφερειακή πτυχή. Ένα τελευταίο ερώτημα. Α, υπάρχει κάποια πρόταση για το ποια είναι η μέθοδος που μπορούν ε, τα κράτη-μέλη να ε, ισορροπήσουν ε, ή να κατανείμουν τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους. Υπάρχει κάποια δική σας έτσι, σκέψη, ας πούμε, αν υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν ας πούμε, να συμφωνήσουν. Δεν θα ήταν καλό και μετά ας πούμε, θα πρέπει να, να αφαιρεθεί ή να καθυστερήσει η χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων, κάποιων projects. Επίσης, ε, έχουμε και μια υπηρεσία η οποία από τον ε, Γενάρη λειτουργεί και το ερώτημα είναι ε, έχει κάποια αρμοδιότητα ώστε να ασχοληθεί με το θέμα των υποδομών. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Τόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει και με μία ερώτηση που έγινε και προηγουμένως. Θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο όλοι να δούμε τα θέματα, να συζητήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο με τους επιτρόπους για την στρατηγική σημασία που θα έχει όλο αυτό το project, όλο αυτό το πρόγραμμα για την ε, προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των επενδύσεων αλλά και της απασχόλησης. Δεν είναι όμως τώρα βέβαια αυτή η στιγμή για να γίνει η αξιολόγηση. Και σε σχέση με αυτά που μας θα ήθελα να πω ιδιαίτερα, ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, προσπάθεια που γίνεται σε προγραμματικό επίπεδο. Ε, υπάρχουν προτεραιότητες, προγραμματικές, ε, ένας σχεδιασμός που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης και, το κανονιστικό, και κανονιστική προσπάθεια σε κανονιστικό επίπεδο που είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι χρειάζεται μια κάποια ρύθμιση σε των, στο τομέα των τηλεπικοινωνιών, και γενικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές, ο προγραμματισμός με πείθουν. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, με πείθει αλλά με ανησυχεί λιγάκι κιόλας η αποτελεσματικότητα αυτού του νέου μηχανισμού. Και αυτό για και η καινοτομία και γιατί μιλάω για, για καινοτομία. Δεν έχω καταλάβει εάν η χρησιμοποίηση των δημοσιονομικών οργάνων που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει ε, εφαρμόζονται με ένα κριτικό βλέμμα. Γιατί δεν ήταν όλες αυτές ε, οι πολιτικές ε, επιτυχημένες. Για, το, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παραδείγματος χάρη το φθινόπωρο του 2008, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά η κρίση, υπήρχε αυτό το ρεκόρ, ένα τότε ένα recover, plan, ένα πλάνο ε, ανόρθωσης και ήταν ε, ε, η δυνατότητα στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων να προσφύγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ήθελα να ρωτήσω ε, τώρα και για, τη δική μου, και για τη δική μου χώρα ε, πόσα χρήματα από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από οπουδήποτε αλλού κατέληξαν τελικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και την κρίση. Λοιπόν, η επαναχρησιμοποίηση σημαίνει να τα χρησιμοποιήσουμε με κριτικό βλέμμα και πολύ ε, προσεκτικά, όχι γενικά να λέμε, λειτουργούν όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτά, τώρα για τα ομόλογα έργου. Εάν είναι πειραματικό, θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, διότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει και το θέμα προσδοκίας. Έχουμε τις ε, ε, εφημερίδες, τις οικονομικές κτλ. που μιλάνε συνέχεια για τα, για τα ομόλογα. Και λέμε τέλος πάντων, γιατί να μην κάνουμε ομόλογα έργου τώρα, που είναι και πολύ πιο εύκολα από τα οικονομικά ομόλογα. Λοιπόν, Τώρα, η ερώτηση που θέλω να κάνω, που την έκανε και, μια, και ένας άλλος συνάδελφος. Αυτά τα ομόλογα έργου, πού βλέπουν να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για μεγάλα έργα τα οποία αυτοχρηματοδοτούνται με τα, μέσω των ομολόγων έργου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πού εμπλέκεται σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι εγγύηση, ε, βοηθάμε να γίνει πιο άμεσα η χρηματοδότηση. Πρέπει να το καταλάβουμε σαφέστερα, διότι αύριο, μεθαύριο, τέλο πάντων κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια μιας αναθεώρησης ή άλλων εργαλείων για τα για, τις, για την διακυβέρνηση μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει πάλι τα ομόλογα έργου και να μας πει τα έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη. Λοιπόν, τα καινοτόμα εργαλεία θέλουμε να, να υπάρχουν και να είναι και επιτυχημένα. Όμως πρέπει να είναι σαφή, διότι μας παρασύρει ο ενθουσιασμός μας και τελικά μπορούμε να καταλήξουμε πουθενά. Μπορεί να ξεκινάμε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά αν το συζητήσουμε και με τις χώρες μας, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη κριτική και όσον αφορά και την βραδύτητα, την βραδύτητα με την οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων και νομίζω πως την έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αμέσως. Ακούστε και όμως και μία ανησυχία για την ε, αυξανόμενη μόχλευση των ε, δημοσίων κονδυλίων και ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ δεν έχει τη δυνατότητα να μοχλευθεί. Γιατί όταν χρησιμοποιεί κανεί κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και αν κατάλαβα καλά τον τοποθετεί ε, στην ε, Τράπεζα Επενδύσεων την Ευρωπαϊκή έτσι ώστε να τα επενδύσει και να ε, δώσει δάνεια, τότε νομίζω πως η ίδια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα έχει τη δυνατότητα να μοχλεύσει τα κονδύλια αυτά και να δανείσει ε, παραπάνω από αυτά τα οποία έλαβε, γιατί έχει το τριπλό α και αυτό γιατί το δανειακό της κεφάλαιο το εγγυώνται τα κράτη-μέλη. Οπότε μπορεί να δανείσει άλλες τράπεζες, ε, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να ακολουθήσει τις κεφαλαιακούς, ε, τους κανόνες περί κεφαλιακής επάρκειας που δεσμεύουν τις άλλες τράπεζες, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία θα της έχει προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Πρώτη ερώτηση, γίνεται αυτό. Και δεύτερο, μας είπατε ότι θέλετε να προωθήσετε τη μακροπρόθεση επένδυση ε, ιδιωτικών κεφαλαίων. Όμως, εμείς και εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να νομοθετήσουμε για, τις, ε, για τα ιδιωτικά κεφάλαια, δηλαδή ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιδοτικά ταμεία, τα οποία τα αποθαρρύνουν από τη μακροπρόθεση επένδυση. Μιλάω για το πακέτο Solvency 2, για τα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάω για τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Είστε λοιπόν σίγουροι πως εμείς οι οποίοι θέλουμε μακροπρόθεσμη επένδυση στις επενδύσεις, δεν είμαστε ήδη οι οποίοι θέτουμε φραγμούς που δεν, ε, που δεν επιτρέπουν σε πολλούς επενδυτές ε, τύπου ταμείων να επενδύσουν. Και έχω και μια τελευταία ερώτηση για κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου δημοφιλές και αυτό είναι η, ε, το θέμα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Πολλές φορές οι επενδύσεις αυτές έχουν σκοπό να αυξήσουν την πιστοληπτική ικανότητα κάποιων δανειστών οι οποίοι δεν έχουν πολύ ψηλά σκορ. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κάποια κράτη ε, έχουν ε, χαμηλή αξιολοπτική ικανότητα. Άρα λοιπόν και τα έργα εκεί ε, θα έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα τους επιτρέψουμε την πρόσβαση στα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λόγω χαμηλής ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης ή θα αλλάξουμε εδώ τους κανόνες ώστε να επιτρέπεται, γιατί υπάρχει το θέμα. Μπορεί να μοχλεύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μπορούμε να ε, τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς να παρακάψουμε τους κανόνες περί περιορισμού κάποιων ταμείων σε επενδύσεις και τρίτον τι γίνεται με την πιστοληπτική ικανότητα ικανότητα και ποιος έχει το τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα δάνεια αυτά από την ΕΤΕ. My question... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημα που έχω να θέσω ακολουθεί το ερώτημα της συναδέλφου Φόρντ για, την, για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Θα υπάρξει ένα ταμείο που θα στοχεύει τα εμπορικώς βιώσιμα επικερδή project και μπορούμε ας πούμε να το συνδέσουμε και με περισσότερα ομόλογα έργο κτλ. Επίσης είπατε ότι περιμένετε ψηλή μόχλευση σε αυτό το ταμείο, 15 με 20%. Αυτό σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν περίπου 50 δις δημόσιο κονδύλι για το Connecting Europe, το συνολικό, η συνολική επένδυση θα φτάσει τα 700, από 752 δις σε ένα αυτό είναι πολύ κοντά στα αμυγός εμπορικά ε, project με τόσο υψηλή μόχλευση η βοήθεια του κρατικού Κορβανά για να ενισχύσει αυτά τα, τα, τα, αυτά τα project δεν είναι και πολύ μεγάλη τελικά. Νομίζετε λοιπόν ότι θα υπάρξει αρκετή ζήτηση για τέτοια ποσά με τέτοιου είδους εργαλεία και δεύτερον, αυτό είναι συμβατό με άλλους τύπους χρηματοδότησης όπως ας πούμε οι επιδοτήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να θέσω άλλο ένα ερώτημα πριν απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Όλοι οι συνάδελφοι είπαν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε υποδομές και χρειαζόμαστε χρήματα, σαφώς. Δεύτερον, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, όπως είπε και η Βίκη Φόρντ, πώς μπορούμε να λάβουμε ιδιωτικό κεφάλαιο που υπάρχει και πώς μπορούμε να το φέρουμε σε τέτοια, ε, ε, σε προγράμματα. Αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να το αποφασίσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά είναι τελικά αυτό που αποφασίζουμε εμείς σε πολιτικό επίπεδο χρήσιμο ή μήπως κάνουμε το αντίθετο. Όποιο επενδύει σε ένα έργο θέλει να, κατα... να έχει και κέρδος, προφανώς. Αλλά αυτό εμείς σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι πάντα ε, συμμορφούμενο με, τον, με την ε, ύπαρξη κέρδους. Και δεύτερον, τα δημόσια κονδύλια που έχουμε είναι περιορισμένα. Πώ θα ε, ε, τεινάξουμε πούμε, το ραβδί και θα γεννηθούν νέα κονδύλια, δεν γίνεται να κάνουμε μαγικά. Ε, εμένα μου δημιουργούνται πολλέ ανησυχίε, πολύ συχνά. Ειδικά σε τέτοιου καιρού τρα, τραπεζικών κρίσεων, α, μου έδειξαν ότι όποιοι λένε ότι θα κουνήσουμε το ραβδί μα και θα γεννηθούν λεφτά, ε, ουσιαστικά είναι άνθρωποι που δίνουν ψευδείς υποσχέσεις. Εγώ έχω μεγάλη ανησυχία για το μήπως κάνουμε τελικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να λύσουμε με ένα μαγικό τρόπο το πρόβλημα των τραπεζών, μήπως προσπαθούμε να το κάνουμε για να λύσουμε και το πρόβλημα των λοιπών κονδυλίων για τα προγράμματα. Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, προφανώς. Πόσο εύκολο, πόσο ασφαλής όμως είναι όλη αυτή η ιστορία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που πρέπει τελικά να απαντήσουμε. Η... Το, το σίγουρο είναι να υπάρξει ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι το μόνο πιο σίγουρο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα και εγώ να έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Λάβατε πολλά ερωτήματα, κάποια μάλλον δεν είναι και εύκολο να απαντηθούν άμεσα. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Θα προσπαθήσω εγώ. Ε, να δώσω λοιπόν μία απάντηση στον κύριο Όντι και στην κυρία της οποίας δεν μπορώ να πω το όνομα. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, τα οποία βεβαίως και θα συγκεντρώσουμε και θα λάβουμε υπόψη τα όσα είπατε και οι δυο σας. Νομίζω ότι μπορώ να πω πως το μέσο αυτό, το εργαλείο αυτό και αυτά τα 50 δις που είναι μεγάλος προϋπολογισμός αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη δική σας ανάλυση, δηλαδή πως ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές. Αυτό είναι βέβαιο και θα πρέπει να δούμε ε, αυτό το οποίο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η φιλοδοξία μας θα πρέπει να συνδυάζεται και με τους δημοσιονομικούς ε, περιορισμούς που έχουμε. Ε, πάντως, την ανάγκη επενδύσεων για την ανάπτυξη θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Τώρα, αν τα ποσά δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά τα οποία διαβάσαμε στα αντίστοιχα της Κίνας, συνδύαση των ΗΠΑ, νομίζω ότι εκτός από το κατά πόσο μπορούμε και σε κινητικό επίπεδο να χτίσουμε αυτές τις υποδομές, γιατί νομίζω ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνδυάζεται και με την εθνική. Μην το ξεχνάτε αυτό όταν μιλάμε για επίπεδο χρηματοδότησης υποδομών. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε πως αυτές οι χρηματοδοτήσεις που προτείνονται στα 50 δις είναι στοχευμένες για να έχουμε ολοκληρωμένες ε, ε, υποδομές, ή εθνικές να ολοκληρωθούν μέσα στα ευρωπαϊκά δίκτυα και ακόμα και αν τα ποσά δεν είναι <coughs> συγκρίσιμα με αυτά τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συγκρίνουμε με αυτά που έχουν άλλα μεγάλα οικονομικά μπλοκ, νομίζω ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά εξαιρετικά ωφέλιμα, γιατί θα κάνουν την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική και το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται κάτω από αυτούς τους τρεις ε, προσανατολισμού και με αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι κατά τη γνώμη μου πολύ φιλόδοξο. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση για την έρευνα που θα καταθέσουμε σε μερικές μέρες. Με ορίζοντα το 2020 ε, θα κάνουμε και κάποιες ε, προτάσεις για το Γαλιλαίο, ε, και για το ε, GMS, τα οποία κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλα, να πρεκοδοτηθούν με υψηλούς προϋπολογισμούς, όχι βέβαια μέσω αυτού του μηχανισμού. Όσο για τις ε, περιφερειακές υποδομές και τις επενδύσεις εκεί, νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα είναι προφανή. Πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε από την εθνική, τις εθνικές επενδύσεις και μετά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα περιφερειακής ε, χρηματοδότησης, γιατί βέβαια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάποια όρια με στα οποία μπορεί να κινηθεί. Το πρώτο στάδιο πάντως το οποίο θα διανύσουμε είναι και το πιο σημαντικό και εδώ θα μεταφέρουμε τα σχόλιά σας ε, στην Επίτροπο μετά από τα όσα ακούσαμε σήμερα. Μιλήσατε για κριτήρια κριτήρια συγκεκριμένα για να γίνουν κάποιες επιλογές έργων ε, και δώσατε και στις μεταφορές ένα παράδειγμα. Όντως είναι κομβικό το θέμα αυτό και η πρότασή μας για τους τρεις κλάδους που συμπεριλαμβάνει ε, βασίζεται σε μια επιλογή ε, έργων που θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη πρωταρχικά την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα φέρουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση και για τις μεταφορές πιο συγκεκριμένα, το δικό σας όραμα, και θα το πω στα αγγλικά, αυτή η συγκέντρωση χρηματοδότησης και σε ε, κέντρα logistics ε, για τις μεταφορές είναι κάτι το οποίο έχουμε εντοπίσει και εμείς όπου ε, χρειαζόμαστε κάποιους κόμβους ε, κόμβους συγκοινωνιακούς που μπορεί να είναι ε, κάποια τέρμιναλ ε, σιδηροδρομικά, μπορεί να είναι κάποιοι λιμένες. Είναι εν πάση σημεία στα οποία θα στηρίξουμε και τις υποδομές αλλά και τη διάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών των logistics τα οποία εκεί θα πρέπει να αναπτυχθούν. Και εδώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα όσα έχουμε στο δικό μας μηχανισμό τις προτάσεις για τα σύνορα της Ευρώπης, της Ευρώπης, εκεί που τα δικά μας δίκτυα συνδέονται με τα μετασυγκοινωνιακά δίκτυα των όμορων χωρών. Έχουμε και τα μέτρα περιφερειακής πολιτικής, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Πάρα πολλά μπορούμε να συμπληρώσουμε. Αύριο στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια σχετική παρουσίαση αλλά και για τους τρεις κλάδους αυτούς θα προσέξουμε ιδιαίτερα τη διάδραση μεταξύ του δικού μας μηχανισμού και της περιφερειακής πολιτικής όχι μόνο σε επίπεδο νομικών διατάξεων που διέπουν τα εργαλεία αυτά, αλλά και στις δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε με τις δικαιούχες χώρες, δηλαδή στις διάφορες εταιρικέ συμφωνίες που θα υπογραφούν και στα επιχειρησιακά προγράμματα και για τους τρεις κλάδους θέλουμε να έχουμε συμπληρωματικότητα μεταξύ του δικού μας μηχανισμού που δίνει την προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία και των όσων κάνουν τα περιφερειακά μέσα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτό αποτελεί δική μας προτεραιότητα. Και δεν είμαι σίγουρος, νομίζω στην ερώτησή σας καλύψατε και το θέμα του Ταμείου Συνοχής και της διαχείρισης αυτού, ε, τα 10 δις τα οποία μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στο δικό μας μηχανισμό, Νομίζω πως αυτό το κομμάτι της δικής μας πρότασης έχει ως σκοπό τις χώρες της συνοχής να τις βοηθήσουν να συγκεντρώσουν τμήμα των επενδύσεων ε, στα σημεία διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία, δηλαδή τα 10 δις ε, θα είναι εστιασμένα και στοχευμένα ε, στα σημεία ε, διαδικτύωσης, αλλά μόνο στις χώρες συνοχής. Είναι λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρίας με, συνολικό, με συνολική πρικοδότηση 10 δις για τα σιδηροδρομικά project που είναι δύσκολα και επίσης για τα οδικά έργα τα οποία είναι διασυνοριακά και επίσης όπου η προετοιμασία είναι δύσκολη. Άρα λοιπόν θα έχουμε χρηματοδότηση με τα ποσοστά των χωρών συνοχής ε, και θα ε, διατηρήσουμε τα ποσοστά αυτά έτσι ώστε ε, το κομβικό δίκτυο που χρειάζεται με αποτελεσματικό τρόπο και αρμονικό τρόπο να συγκροτηθεί επιτέλους και στις χώρες της συνοχής. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις που άκουσα, που είναι τα καινοτόμα μέσα εργαλεία χρηματοδότησης και την ΕΤΕ, νομίζω πως ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν κάτι να σχολιάσουν. Ακόμα και κάτι διαφορετικό. Διαφορετικά μπορούμε να κλείσουμε με τα, εργα... με τα εργαλεία χρηματοδότησης. Δύο ερωτήσεις ετέθησαν για την ενέργεια. Το ένα είναι για την πρόταση για την χορήγηση αδειών θεωρούμε ότι όντω είναι φιλόδοξο μεν, ρεαλιστικό δε. Καταρχάς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι άδειε ε, υπάρχουν όταν ε, πρέπει να γίνουν οι επενδύσει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2020 για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις. Για τα τρία χρόνια είναι υποχρεωτικά όπως προτείνεται, είναι η μέγιστη προθεσμία, αλλά η πρόταση επίσης περιέχει και διάφορα εργαλεία, τα οποία θα εξασφαλίσουν ε, την, τον σεβασμό της προθεσμίας των τριών ετών. Όπως σας είπα, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, είναι μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σήμερα σε κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, παραδείγματος χάρη, ή της Δανίας, της Ιρλανδίας, των κάτω χωρών και πρόσφατα και στην Γερμανία ισχύει η προθεσμία αυτή, άρα είναι ε, εφικτή. Η πρότασή μας αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, τώρα, τι θα γίνει εάν η αρμόδια αρχή δεν πάρει μια απόφαση για το κατά πόσον θα πρέπει να δώσει την άδεια στην προθεσμία αυτή των τριών ετών. Οι κυρώσεις είναι οι φυσιολογικές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική. Η Κομισιόν θα αντιδράσει. Όμως πριν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνουμε στην πρόταση μας είναι και πολύ αυστηρός έλεγχος της εφαρμογής των project σε περιφερειακή βάση ε, όπου ε, οι επιχειρήσεις, οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις, ε, οι υπεύθυνοι και οι συμμετέχοντες στο όλο project θα ε, συναντώνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν και να συζητάνε τα προβλήματα, τα εμπόδια κτλ. έτσι ώστε να αναλυφθεί δράση και να διορθωθεί η κατάσταση πριν να περάσουν τα τρία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την ε, υπηρεσία ή τον οργανισμό, ο οποίος ε, δημιουργήθηκε στις αρχές του χρόνου και έχει την έδρα του στην Λουμπλιάνα, εκεί θα παίξουν ένα ε, σοβαρό ρόλο αυτή η οργανισμός και όσον αφορά το, την ρύθμιση αλλά και την παρακολούθηση και τον έλεγχο έτσι ώστε να εφαρμοστούν έγκαιρα τα project. Να πω δύο λόγια για την συμπληρωματικότητα και την χρηματοδότηση που θα υποβληθεί μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής. Όσον αφορά την, τις επενδύσεις αυτές καθεαυτές, θεωρούμε ότι τα χρήματα αυτά θα έχουν έναν έντονο συμπληρωματικό χαρακτήρα. Βέβαια, θεωρούμε ότι τα ταμεία συνοχής ε, θα είναι πιο ε, ελκυστικά εφόσον υπάρχουν τα χρήματα από το Ταμείο Συνοχής. Ε, υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίε μας ε, δυνατότητα και για περαιτέρω ρευστότητα με την πρόσβαση σε άλλα χρηματικά, χρηματοδοτικά εργαλεία. Η συνθήκη αναφέρεται και σε ένα άλλο είδος συνοχής έτσι ώστε οι πιο απομακρυσμένες περιοχές να προσεγγίσουν το κέντρο μέσω έργων υποδομής και δίδεται μία κάπως διαφορετική απάντηση από αυτή που δίνουν τα, τα το Ταμείο Συνοχής. Υπάρχει βέβαια και το ψηφιακό κάσμα, το ε, ψηφιακό χάσμα το οποίο δεν αναφέρεται στην ε, συνθήκη, διότι τότε δεν υπήρχε ψηφιακό χάσμα. Αλλά και αυτό αντιμετωπίζεται τώρα. Okay, let me try να προσπαθήσω κι εγώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο βαθμό που μπορώ. Υπήρξαν αρκετά ερωτήματα για το ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι η μηχανική όλων αυτών των, αυτού του προγράμματος, μάλλον των ομολόγων έργων. Η συνάδελφος εδώ πάνω στο βήμα είπε ότι όντως είναι ανάληψη μεικτή ε, του κινδύνου είναι μάλλον πιο έμεσος ο τρόπος του να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε μέσω ε, ε από κοινού ανάληψης των, των κινδύνων παρά με τη χρήση άμεσων εργαλείων που είναι μερικές φορές πιο δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε σαφή όρια στην, στο ποσοστό ευθύνης ας πούμε. Μπορεί βέβαια να πείτε γιατί συμβάλλει η Κομισιόν. Δεν θα πρέπει να είναι η Τράπεζα Επενδύσεων που τα κάνει αυτά από μόνη της. Όπως σωστά είπατε υπάρχουν ε, ανησυχίες για την αμόχλευση των ε, τραπεζών. Και αυτό που προτείνουμε εμείς με αυτό, αυτή την πρωτοβουλία των ομολόγων ε, έργων είναι ότι ναι, εντάξει, από, την, ε, από τη μία είναι πιο επικίνδυνο από, το απλό, από τον απλό δανεισμό από την ε, τράπεζα, αλλά κυρίως μιλούμε για μικρό, ε, μικρό κόστος για, για τη χρηματοδότηση των έργων, ας πούμε ένα 20%, ενώ σε, μια, σε ένα απλό δανεισμό μπορεί να φτάσουμε το 50%. Το αποτέλεσμα του να αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο η Κομισιόν και, η, και που δανείζει λιγότερα και της κατανομής των αρμοδιοτήτων είναι ότι δεν θα υπάρχει αύξηση, καθαρή αύξηση της, μόχλησης, της μόχλευσης από την τράπεζα. Άρα, η τράπεζα θα μπορεί να διατηρήσει και την αξιολόγησή της και δεν θα αναλάβει τεράστιο κίνδυνο. Βεβαίως, μετά μπορεί κάποιος να πει ναι αλλά αυτό δεν μετακυλεί το πρόβλημα στην τράπεζα. Ε, ναι, αλλά αυτό είναι δουλειά και της Κομισιόν, να εξασφαλίσει δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποιες συνετές παράμετροι τις οποίες πρέπει να τηρεί η τράπεζα. Και γενικώ ε, η τράπεζα και οι διεθνείς ε, οργανισμοί είναι πολύ συντηρητικά ιδρύματα, ίσως πολύ συντηρητικά για κάποιους αλλά για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θεσμικό όργανο, όπως λέει η συνθήκη. Και εμείς ως θεσμικά όργανα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες να ελέγξουμε ή να ζητήσουμε από την τράπεζα να μας πει τι κάνει από, ό,τι, από όσο θα μπορούσαν να το κάνουν κάποιοι άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη όταν ρωτάτε γιατί χρειάζονται οι άλλοι εταίροι πλην της ε, ΕΤΕ. Αν θέλουμε να έχουμε εμπειρογνωμοσύνη ε, και γεωγραφική κάλυψη για κάποιους τομείς και τη μεγαλύτερη δυνατή εφαρμογή των στρατηγικών μας, προφανώς χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερους εταίρους. Βεβαίως, Επίσης ισχύει ότι κάποιες από τις άλλες τράπεζες, ε, οι τράπεζες οι επενδυτικές γενικώ, η Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουν και αυτές τους περιορισμούς τους σε ό,τι αφορά το καταστατικό τους. Και βεβαίως έχουμε δεσμευτεί να δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα άλλων τέρων που θα χρηματοδοτήσουν. Θα, συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση πλατφόρμα για όλους, γιατί κάθε, κάθε τράπεζα έχει τους δικούς της περιορισμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ρυθμιστικά στοιχεία. Γνωρίζουμε τις, ε, τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το ε, Φεργκιότητα 2 και άλλες προτάσεις, αλλά έχουμε τελικά διαφορετικές αντιλήψεις στα κράτη-μέλη απέναντι σε αυτές τις, ε, τα ρυθμιστικά εργαλεία. Άλλοι λένε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, άλλοι λένε ότι δεν ανησυχούν τόσο πολύ, γιατί μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας προσέγγιση και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, στις συζητήσεις λοιπόν που κάνουμε με άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να δούμε πού είναι τελικά το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, που, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος εφαρμογής, ανακράτος μέλος των διαφόρων κανονισμών. Αυτό θα συνεχίσουμε να το Ψάχνουμε. Και σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλή αξιολόγηση, που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθόλου τα χρηματοδοτικά εργαλεία ή τα ομόλογα, όντως και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το, να το δούμε. πολλές φορές η προσέγγιση των ε, οίκων αξιολόγηση είναι αρκετά δογματική, αλλά μέσω των ομολόγων ε, έργων είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε ε, προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την ε, αξιοπιστία του κάθε κράτους μέλους. Βεβαίω λαμβάνονται υπόψη και οι κίνδυνοι που υπάρχουν στη χώρα αυτή που θα αναλάβει το έργο. και για το αν μπορούμε, αν υπάρχει τρόπος, να ξεπεράσουμε το όριο που έχει τεθεί για την κάθε χώρα, που συνήθως ε, είναι όριο που υπάρχει για οποιοδήποτε φορέα ασχολείται με το έργο στη χώρα αυτή, ε, θα πρέπει και αυτό να το, να το δούμε. Μπορεί να είναι θέμα δηλαδή σχεδιασμού για να μπορέσουμε να το λύσουμε καλύτερα το πρόβλημα και θέλουμε όντως να το λύσουμε και στα πλαίσια της πιλωτικής φάσης. Νομίζω ότι έχω απαντήσει έτσι γενικώ. Σύντομα να πω δύο λόγια, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στα γρήγορα απλώς να επαναλάβω πως ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ένα κομμάτι από το μηχάνισμα αυτό θα μεταφέρεται από τον προϋπολογισμό στους ε, χρηματοσπιστικούς οργανισμούς που θα έχουν αναλάβει το κομμάτι των εγγυήσεων, άρα λοιπόν δεν κινδυνεύει ο προϋπολογισμός και για την ΕΤΕ η απόφαση για τα έργα θα γίνεται από τις τράπεζες, θα παίρνεται από τις τράπεζες και βεβαίως ε, σε αυτά τα εργαλεία καταμερισμού κινδύνου θα λαμβάνει υπόψη τις ίδιες τις, τις δανειακές υποχρεώσεις και το κεφάλαιό της έτσι ώστε να μην κληθεί να ξεπεράσει τα όσα ορίζει νομοθεσία. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε είναι μια καλή γεωγραφική κατανομή έτσι ώστε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και οι επενδυτές να ε, κάνουν ένα διάλογο που θα προετοιμάσει τα κατάλληλα έργα, τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα είναι μόνο καλά έργα, αλλά θα είναι ε, και διασπαρμένα στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο για τα ομόλογα έργο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ε, ε, έναν συνδυασμό μεταξύ των κανόνων χρηματοδότησης αλλά και των κανόνων και των θεμάτων που μας απασχολούν επί τόπου, έτσι ώστε ε, να, μην να μην συγκεντρώσουμε τα projects ε, σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά να τα διασπείρουμε σε όλες τις περιοχές γεωγραφικού ενδιαφέροντος. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους της Κομισιόν για όλες αυτές τις πληροφορίες. Είμαι ευγνώμων που δεν επικεντρωθήκαμε μόνο σε επιμέρους ε, projects και μιλήσαμε γενικώ το ότι περισσότερες, χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις ε, για τις υποδομές, για την ενέργεια, για την κοινωνία των πληροφοριών, για τις μεταφορές, είναι σαφές. Το ξέρουμε όλοι και χαίρομαι που οι συνάδελφοι ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν για τα εργαλεία που υπάρχουν ή για την ελπίδα που υπάρχει για ύπαρξη νέων ε, εργαλείων, αν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ε, πιθανό πρόβλημα, γιατί αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Η, αυτή η φαντασία οι προσδοκίε που δημιουργούνται κάθε φορά ε, μπορεί να μα οδηγήσει τελικά σε πολλά προβλήματα. Οπότε χαίρομαι που ετέθησαν αυτά τα ερωτήματα στην Κομισιόν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αν υπάρχει ε, σαφέ πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να λειτουργήσει και κατά πόσο τελικά χρησιμοποιούμε το εργαλείο που έχουμε του, των ιδιωτικών επενδύσεων. Γιατί εκεί υπάρχει το κεφάλαιο. Και ε, βεβαίω αυτό θα ήταν και ο πιο εύκολος και ο πιο άμεσος τρόπος για να είμαστε και ε, πιο φιλική ε, ω προ τι υποδομέ ό,τι αφορά τι επενδύσει και να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτή την δημιουργικότητα που μα ε, διαπνέει. Θα συνεχίσουμε να το συζητούμε το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά ουσιώδου σημασία. Χαίρομαι που ήσασταν εδώ μαζί μα σήμερα. Χαίρομαι που μα απαντήσετε σε έναν πρώτο γύρο ερωτήσεων και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, να πάμε στο επόμενο σημείο. Δεν με ακούει κανένα όμω. Τι έγινε ακριβώ και συζητάτε όλοι μεταξύ σα σε πηγαδάκια. Um Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαστε στην αγορά, ούτε σε συνεδρίαση επιτροπής. Ε, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε έξω να συζητήσετε, αν μιλάτε για κάτι άσχετο με το θέμα μας. Ladies and Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Επόμενο σημείο. Μα πρέπει να ξεκινήσουμε. Mr. Klaus Forel Ο κύριος Klaus Φορέλ Πέτερσεν είναι εδώ. Αν θέλετε καθίστε. Yeah. Because time is money. Okay. And we have... Ο χρόνος είναι χρήμα και χρήματα δεν έχουμε.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 Λοιπόν, ε, ελπίζω οι υπόλοιποι συνάδελφοι να καθίσανε για να συνεχίσουμε. Το πρόβλημα που είχαμε το πρωί το έχουμε και τώρα. Για κάποιο λόγο τα κομπιούτερ και, τα, και, το προτζέκτορας δεν, ε, δεν συνδυάζονται, δεν συνεργάζονται και προφανώς δεν μπορούμε και να δουλέψουμε χωρίς όλη αυτή την τεχνολογία. Να περιμένουμε κανένα δυο λεπτά και αν δεν ε, τα καταφέρουμε να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση. Λοιπόν, συνάδελφοι, ξεκινούμε. Θα δούμε μια μελέτη για τα προβλήματα, για τα εμπόδια και τις βέλτιστες πρακτικές για την δοκιμή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για τα καλά. Μάλλον βέβαια έτσι όπως είναι ο τίτλος μάλλον θα μιλήσουμε για τα άσχημα πρώτα και θα αφήσουμε τα καλά για το τέλος. Έχουν μείνει λίγοι συνάδελφοι. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Economic. And then you can start if you want. Και αν θέλετε μπορείτε και να ξεκινήσετε. Αλλά χρησιμοποιήστε αυτό το μικρόφωνο γιατί αλλιώς δεν θα σας ακούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω και να σας πω για την δουλειά που έχουμε κάνει. Ε, είμαι στην Κοπενχάγη, ασχολούμαι με τα οικονομικά και εκεί στο Πανεπιστήμιο κάναμε μια μελέτη για σας για το πώς αυτή η δοκιμή των ΜΜΕ μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη και στις υπηρεσίες της Κομισιόν. Όπως ξέρετε, η δοκιμή ΜΜΕ είναι ένα κομμάτι της, ε, των δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το 2008 γιατί ε, η Κομισιόν είπε ότι θα εφαρμόσει αυτή την δοκιμή και τα κράτη ε, από τα κράτη-μέλη ζητάμε να εφαρμόσουν αυτή την δοκιμή όταν υποβάλλουν νέες προτάσεις. Αυτή η δοκιμή, δοκιμή ε, ελέγχει, αν θέλετε, τον αντίκτυπο και τις συνέπειες των νομοθετικών προτάσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που κάναμε είναι να δούμε κατά πόσον αυτό, αυτό το, αυτή η δοκιμή των συνεπειών στις, ε, στα ΜΜΕ, στις ΜΜΕ χρησιμοποιείται, ε, εάν χρησιμοποιείται, πώς χρησιμοποιείται, τι εμπόδια υπάρχουν εάν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν εφαρμόσουν αυτή την δοκιμή, ποια, εάν υπάρχουν καλά παραδείγματα χρήσης αυτού, αυτής της δοκιμής. Στηρίξαμε τη μελέτη μας σε δύο πράγματα. Μία έρευνα που έκανε η Κομισιόν μια έρευνα όπου όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν υπεύθυνα για την δοκιμή των ΜΜΕ ή παρόμοια δοκιμή ε, απήντησαν ε, σε ένα ερωτηματολόγιο. Είχαμε τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων από τις 27 χώρες μέλη. Μετά κάναμε σε 7 κράτη-μέλη μια, ε, την έρευνα κάποιων περιπτώσεων. Η Αυστρία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Λετωνία συμμετείχαν σε αυτές τις ε, έρευνες των ε, συγκεκριμένων περιπτώσεων. Τι θα κάνουμε τώρα. Ε, έχουμε και την διαφάνεια. Θα σας ε, παρουσιάσω καταρχάς ε, τα βασικά μηνύματα. Μετά θα μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιείται η δοκιμή αυτή στα κράτη-μέλη και από την Κομισιό. Μετά θα σας μιλήσω για τα εμπόδια τα οποία συναντήσαμε και μετά θα αναφερθώ στις συστάσεις τις οποίες θα θέλαμε να υποβάλουμε και σε εσά και στην Κομισιό και μετά θα υπάρχει και χρόνος για ερωτήσεις και ελπίζω και για απαντήσεις. Τώρα τα βασικά μας μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι δεν εντυπωσιαστήκαμε από το εύρος χρησιμοποίησης της δοκιμής αυτής στα κράτη-μέλη. Και στα κράτη-μέλη αλλά και στην Κομισιόν. Μόνο 15 κράτη-μέλη και οι, Ευρωπαϊκές, οι επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιούν τη δοκιμή ΜΜΕ ή παρόμοιες δοκιμές και αυτό όμως σε επίπεδο ad hoc σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και στα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν την δοκιμή με κάπως πιο οργανωμένο τρόπο και πιο συστηματικά οι υπηρεσίε τη ε, Κομισιόν χρησιμοποιούν την δοκιμή αυτή στι περισσότερε των περιπτώσεων, αλλά και εκεί που εφαρμόζεται το, η δοκιμή δεν γίνεται με έναν οργανωμένο τρόπο. Άρα με όλα αυτά τα στοιχεία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση ε, ε, της χρησιμοποίησης των δοκιμών, κυρίω σε επίπεδο κρατών μελών. Δεύτερον, η έρευνα μας αποδεικνύει ότι υπάρχουν κάποιες βασικές προκλήσεις για το πόσο μπορεί να εφαρμοστεί η δοκιμή αυτή και αυτό το, στο, στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε λέει ότι μία σειρά κατευθυντηρίων γραμμών δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη δεν ταιριάζουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορετικές προκλήσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Και μέσω της μελέτης και μέσω των απαντήσεων που πήραμε, ε, είδαμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που πρέπει να εφαρμόσουν καταρχάς κάποιες βασικές πολιτικές, Δηλαδή πρέπει να δούνε ποιες είναι οι πολιτικές ε, που πρέπει να εφαρμόσουν για να ε, μπορέσουν να εφαρμόσουν την δοκιμή ΜΜΕ. Θα πρέπει δηλαδή καταρχάς να υιοθετήσουν κάποιες πολιτικές θέσεις και μετά να εφαρμόσουν τη δοκιμή. Περισσότερα, τα περισσότερα κρατημέλη δεν έχουν καν υιοθετήσει αυτές τις πολιτικές θέσεις. Μετά υπάρχει και άλλη μια ομάδα κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει κάποιες πολιτικές θέσεις και έχουν εφαρμόσει και κάποιες ε, διαδικασίες, έχουν ε, αποφασίσει την δοκιμή ΜΜΕ, όμως εκεί δεν υπάρχει συστηματικότητα. Δηλαδή, σε κάποιες μόνο περιπτώσεις η δοκιμή ΜΜΕ γίνεται. Δηλαδή, σε λίγες περιπτώσεις ε, αξιολογείται η συνέπεια των νέων νομοθετικών προτάσεων στις, στα, στις ΜΜΕ. Επίσης, έχουμε και χώρες όπου χρησιμοποιείται η δοκιμή με σωστό τρόπο και υπάρχει ένας προηγμένος τρόπος για τη χρησιμοποίηση της δοκιμής, αλλά και εδώ ακόμα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε διαφορετικό επίπεδο μεν, αλλά υπάρχει και η πρόκληση της συμμόρφωσης εδώ. Δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις πλέον προωθημένες και προηγμένες μεθόδους σε όλες, σε τις περιπτώσεις. Τι συστήνουμε ε, μέσω της μελέτης μας. Καταρχάς ε, ότι η εφαρμογή θα πρέπει να προχωρήσει, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, δηλαδή υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να βάλουν κάποια τάξη πρώτα, σε άλλα μπορεί ε, να, χρειάζεται να εφαρμόσουν μια πιο προηγμένη μέθοδο για να βελτιώσουν τα, όσα ήδη εφαρμόζουν. Μετά ίσως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η δοκιμή και να υιοθετηθούν κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο την πολιτική, χρειάζεται να έχουμε και κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να υλοποιηθεί η δοκιμή. Τρίτον, πρέπει να υποστηρίξουμε την εφαρμογή. Δηλαδή χρειάζομαστε και κάποια μέτρα ελέγχου στα κράτη-μέλη, όπως υπάρχουν στην Κομισιόν παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή την δοκιμή, θα πρέπει να έχουν την εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία, θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα help desk, να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δοκιμών αυτών. Και η τελευταία σύσταση, και θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, είναι το τεστ, έτσι όπως το βλέπουμε το η δοκιμή, έτσι όπως την βλέπουμε τώρα, είναι ένα κομμάτι ενός γενικότερου συστήματος για να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Άρα δεν θα πρέπει το, η δοκιμή αυτή να είναι αυτόνομη, ε, θα πρέπει να αποτελεί ένα κομμάτι ενός γενικότερου συστήματος. Ε, πιστεύουμε ότι η δοκιμή των, ε, ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελέσει ένα κομμάτι μιας, ενός γενικότερου συστήματος ε, ελέγχου, αν θέλετε, και αποτίμησης των καταστάσεων. Θα σας πω λίγο πολύ τι είναι αυτό το, αυτή η δοκιμή, τι είναι αυτό το τεστ. Ο ορισμός που δίνει η Κομισιό και που εφαρμόζουν και κάποια κράτη-μέλη είναι ότι είναι μια διαδικασία με μάλλον αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που έχει τέσσερα στάδια. Θα πρέπει καταρχάς να αρθείτε σε επαφή με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να έχεις το απαραίτητο feedback για το πώς οι νέες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου θα τις επηρεάσουν. Πρέπει να γίνει μια προκαταρκτική αξιολόγηση, κατά πόσον θα ε, η νομοθεσία αυτή θα επηρεάσει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή κάποιες από αυτές. Τρίτον, θα πρέπει να γίνει μια μέτρηση του αντικτύπου, άρα θα πρέπει να ποσοτικοποιήσεις, αν θέλετε, ε, το οικονομικό κόστος, το διοικητικό κόστος, πώς θα ε, επηρεάσει την ανταγωνιστική θέση της, της επιχείρησης αυτής όταν θα εφαρμοστεί αυτή η νέα νομοθεσία. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητήσουμε μιλήσουμε, να ρωτήσουμε τις ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν θα μπορούσαν να καταλήξουν στον ίδιο στόχο εφαρμόζοντας διαφορετικά μέτρα, δηλαδή θα πρέπει να δούμε μήπως, τι, μέτρα χρειάζονται αν μπορεί να, έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση, μια αντιστάθμιση, μια αποζημίωση που θα τις βοηθούσε να εφαρμόσουν καλύτερα την νομοθεσία. Ένα σωστό εφαρμοσμένο τεστ μπορεί να βοηθήσει τους, νομοθέτες, τους νομοθέτες διότι θα μπορέσουν να δούνε ποιους θα επηρεάσουν η νομοθεσία αυτή. Ε, μπορεί οι νομοθέτες να πετύχουν τη σωστή ισορροπία, ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, σε ποιο βαθμό και πόσο θα βοηθήσει τους αποδέκτες της. Και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε έναν καλύτερο κανονισμό δηλαδή. Δηλαδή θα υπάρχει καλύτερη ποιότητα του νομοθετικού έργου. Και αυτό προσπαθεί να βοηθήσει και αυτή η δοκιμή, αυτό το τεστ. Τι δείξαμε στην έκθεσή μας με βάση τις απαντήσεις που πήραμε από τα 27 κράτη-μέλη είναι ότι 21 κράτη-μέλη μας λένε ότι η χρήση του, της δοκιμής ε, γίνεται, όμως αν τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά, λιγότερα κράτη-μέλη από αυτά, από τα 21 ε, το εφαρμόσουν. 15 κράτη-μέλη λένε ότι το χρησιμοποιούν το τεστ αυτό πάντα ή στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν ε, προετοιμάζεται ε, η νέα προετοιμαζεται η νεα νομοθεσια και όταν τις ρωτήσαμε όμως πόσες δοκιμές έκαναν το 2010, είδαμε ότι σε 11 κρατημέλη έγιναν 20 δοκιμές όλες και όλες. Εάν λέτε ότι κάνετε πάντοτε τη δοκιμή αυτή, δεν είναι, δεν μπορεί να, δεν είναι αξιόπιστο, αξιόπιστη απάντηση 20 δοκιμές το χρόνο. Επομένως, Έχουμε 15 κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τη δοκιμή, 6 κράτη-μέλη που σπάνια την εφαρμόζουν και άλλα 6 τα οποία δεν τη χρησιμοποιούν. Αυτό το οποίο εντοπίσαμε επίσης είναι κατά πόσον υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που ε, βοηθάνε τις κυβερνητικές ε, υπηρεσίες να εφαρμόζουν το, τη δοκιμή αυτή. Τι βρήκαμε. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, σε διαφορετικό βαθμό υπάρχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι σε αποκεντρωμένες ε, ε, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες ε, εφαρμόζουν τη δοκιμή αυτή και κάθε υπηρεσία την εφαρμόζει με τον δικό της τρόπο. Και αυτό ισχύει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Επομένω, έστω και αν υπάρχουν κάποιε γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ, ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η δοκιμή ποικίλει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια όλων αυτών για το, πώς, το πόσο εφαρμόζεται και εκτελείται η δοκιμή ποικίλει στα, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Έστω και επομένως ε, Μάλλον 12 κράτη-μέλη λένε ότι έχουν εκφράσει ποσοτικά τις συνέπειες τα αποτελέσματα. Όντως είναι ζωτική σημασία να εκφράσετε ποσοτικά τις απαντήσεις αν θέλετε και τις, αποτελέσματα της δοκιμής έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μια ε, νομοθεσία επηρεάζει αρνητικά ή όχι τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 16 κρατημέλη λένε ότι λόγω ακριβώς των αποτελεσμάτων της δοκιμής κάπως μετριάζουν αν θέλετε την ε, νέα νομοθεσία για να μην υποστούν ε, βλάβη ή ζημιά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα το πόσο συχνά ή πόσο σπάνια εφαρμόζουν την δοκιμή ε, και πώς την ε, εφαρμόζουν τη δοκιμή εξαρτάται από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Πρέπει να υπάρχουν και βέβαια και συγκεκριμένα εργαλεία για να γίνεται σωστή η... σωστά, με σωστό τρόπο η δοκιμή. Τέλος πάντων, η γενικότερη ιδέα, η σφαιρικότερη ιδέα εμφανίζεται σε αυτή τη διαφάνεια. Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα που είχαμε, αναλύοντας τα κράτη-μέλη με βάση δύο διαστάσεις, δηλαδή κατά πόσο χρησιμοποιούν συστηματικά την δοκιμή ή χρησιμοποιούν πιο προηγμένα μέσα και μεθόδους και έχουμε δύο ομάδες. Έχουμε μια προχωρημένη ομάδα κρατών μελών όπου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Δανία, παραδείγματος χάρη. Και στην άλλη πλευρά έχουμε τους ε, αρχάριους που είναι η Πορτογαλία, η Ιταλία, η, Ιστανή, η Εστονία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Σλοβενία και στο ενδιάμεσο έχουμε τους οπαδούς αν θέλετε, αυτούς που ακολουθούν οι προηγμένες χώρες, η, προηγμένη ομάδα αν θέλετε μάλλον, ε, χρησιμοποιούν και προηγμένες μεθόδους ε, και ε, εφαρμόζουν συστηματικά τη δοκιμή. Οι αρχάροι ακόμα δεν έχουν υιοθετήσει τις πολιτικές θέσεις που είναι απαραίτητες και σπάνια χρησιμοποιούν τη δοκιμή και οι ενδιάμεσοι αν θέλετε, οι αυτοί που ακολουθούν, έχουμε κάποιες χώρες που χρησιμοποιούν συστηματικά τη δοκιμή, αλλά έχουμε και κάποιες χώρες που το χρησιμοποιούν ε, σπάνια. Αυτή είναι η ευρύτερη εικόνα επομένως. Τώρα, η Κομισιό που τοποθετείται, γιατί και οι υπηρεσίες της Κομισιό απήντησαν ε, στο, στο ερωτηματολόγιο, ε, θα τους τοποθετούσαμε στους προχωρημένους. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα όμως τώρα. Ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν αυτές οι, οι, ομάδες των χωρών μελών. Για τους αρχάριους, όπως σας είπα, είναι ζωτική σημασία να υιοθετηθεί μια πολιτική θέση επί του θέματος. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι χώρες αυτές ε, ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν νέα νομοθεσία, θα πρέπει μάλλον όταν εφαρμόζουν νέα νομοθεσία να εφαρμόζουν και τη δοκιμή. Αυτό είναι βασικό. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουν την δοκιμή αυτή μέσω κάποιας δομής. Δηλαδή κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνο ε, και υπόλογος για την, για την δοκιμή αυτή. Είναι βασικό αυτό και σημαντικό αν θέλουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Και αυτέ είναι βασικέ προκλήσει. Εάν δεν εφαρμόζονται αυτά τα θέματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στου στους ενδιάμεσου τώρα, στην ενδιάμεση ομάδα, υπάρχουν κάποιε ασυνέπειε. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική θέση, α όμω δεν χρησιμοποιείται συστηματικά το τεστ. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίε που πρέπει να εφαρμόζουν οι κυβερνητικέ αρχέ, οι κυβερνητικέ υπηρεσίε για την εκτέλεση της δοκιμής. Το βασικό εμπόδιο τώρα στις προηγμένες χώρες είναι η έλλειψη συμμόρφωσης. Δηλαδή, υπάρχει η δοκιμή, έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται συστηματικά, όμως δεν υπάρχει συμμόρφωση. Παραδείγματο χάρη η έκφραση ποσοτικά των αποτελεσμάτων της ε, δοκιμής. Τι είπαμε όταν ήρθαμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη και με τις ε, ενώσεις επαγγελματικές, στην ομάδα των αρχαρίων Ιταλία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες ε, ήταν ε, οι συνομιλητές μας ε, και από αυτά που ακούσαμε από την Ιταλία είδαμε ότι δεν υπάρχει δέσμευση, από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να εκτελέσουν τη δοκιμή αυτή. Στην Ρουμανία μας είπαν ότι η δομή που απαιτείται για την εφαρμογή της δοκιμής δεν υπάρχει. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για αυτές τις χώρες. Σαφής η έλλειψη. Στην ομάδα των μεσαίων το βασικό είναι πώς χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές. Στη Λετωνία για παράδειγμα μας είπαν πως πολλές φορές είναι δύσκολο οι δημόσιοι υπάλληλοι από δυσκολο η δημόσια υπουργεία που δεν ε, εργάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών να κάνουν αυτές τις δοκιμές. Τα υπόλοιπα Υπουργεία δεν καταλαβαίνουν τι προσφέρουν οι δοκιμές αυτές. Είναι μια πρόκληση λοιπόν και όταν θέλει κανείς να τις εφαρμόσει ε, οριζόντια σε όλα τα Υπουργεία είναι δύσκολο οι άλλοι κυβερνητικοί φορείς και τα Υπουργεία να τα εφαρμόσουν, μια και δεν ε, αισθάνονται πως λειτουργούν, δεν το πιστεύουν, δεν ξέρουν τι αποτελέσματα δίνει. Στην Αυστρία είναι τα βιομηχανικά επιμελητήρια και ενώσει που επέκριναν και είπαν πολλές φορές το κάνουν οι κυβερνήσεις ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Και το πώς αποφάσισαν βέβαια ότι δεν χρειάζεται αυτή η δοκιμή, τι να σας πω. Ε, μάλλον κάναν βουντού. Άρα λοιπόν αυτό που διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται και πολιτική βούληση από τις κυβερνήσεις, όχι μόνο από τις διοικήσεις, γιατί αν υπάρχει οι κατευθυντήρες γραμμές μετασυντάσσονται. Στην προχωρημένη ομάδα των ε, κρατών μελών, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία, δύο κράτη τα οποία κάνουν αρκετά προωθημένες δοκιμές, μας είπαν τα εξής στη Δανία μας είπαν οι κατευθυντήριες γραμμές είναι καλές, αλλά τα Υπουργεία έχουν και ένα βαθμό αυτονομίας, άρα λοιπόν Αυτό φαίνεται και από τις δοκιμές γιατί δεν έχουν όλες την ίδια ποιότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί πρόβλημα συμμόρφωσης με κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ενδεχομένως επομένως του να είναι άριστες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει μερικά από τα πιο προχωρημένα συστήματα ακούσαμε επικριτικά σχόλια γιατί βέβαια όλα τα Υπουργεία δεν συμμορφώνονται με τον ίδιο τρόπο. the European Commission. Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε ποιες είναι οι βασικές μας παρατηρήσεις. Σίγουρα από τις ε, μελέτες που κάναμε πιστεύουμε πως έχουμε προχωρήσει και θεωρούμε πως οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα απερίφραστο τμήμα των ε, κατευθυντήριων γραμμών για τον οικονομικό αντίκτυπο και γίνεται και με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και μάλιστα ε, είχαμε και κάποιες πειθαρχικές συνέπειες ε, από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δοκιμές. Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται ιδιαίτερα προωθημένα και προχωρημένα συστήματα. Διαπιστύνουμε όμως από τις εκθέσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο που διαβάσαμε πως το περιεχόμενο αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ε, κατευθυντές γραμμές, οι μεμονωμένες υπηρεσίες αποφασίζουν οι ίδιες για το πώς θα τις διεξάγουν. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται κατά περίπτωση. Με αποτέλεσμα το περιεχόμενο και, το, και η ποιότητα αυτών των δοκιμών να διαφέρει. Κάτι που διαπιστώσαμε επίσης είναι να λείπουν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ίδιες ε, τις δοκιμές, για το πώς έχουν στηθεί στην έκθεση για την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου. Δηλαδή σε ποιο βαθμό έγινε η δοκιμασία και ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτά δεν βρίσκουμε. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι δοκιμές ε, αυτές είναι διαφορετικής, ποιότητα ποιότητας από γενική διεύθυνση σε γενική διεύθυνση. Από τη γενική διεύθυνση επιχειρήσεων σχολίασαν ε, το εξή πως υπάρχουν ε, διάφορες υπηρεσίες οι οποίες έχουν διαφορετική ευαισθησία για το θέμα. Αυτό μας είπε ο αξιωματούχος από τον οποίο πήραμε συνέντευξη και η βιομηχα... η... τα βιομηχανικά και επιχειρηματικά επι... μελητήρια μας είπαν πως αποτελούν έναν ε, κατάλογο, ένα ευχολόγιο ε, από όπου επιλέγουν οι γενικές διευθύνσεις ό,τι προτιμούν να κάνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι λοιπόν ένα κλειστό κουτί ε, το οποίο όταν ανοίγουμε βρίσκουμε να λείπουν στοιχεία, στοιχεία συνδετικά. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο για τον αναγνώστη μια έκθεση αξιολόγηση οικονομικού αντίκτυπου να δει ποια η δοκιμή έγινε, ποιο είναι το περιεχόμενό τη και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτή. Ω τμήμα τη μελέτη, εξετάσαμε 22 με συγχωρείτε, εκθέσει οικονομικού αντίκτυπου από διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει και βρήκαμε και βρήκαμε λοιπόν πως μόνο σε μία μειοψηφία περιπτώσεων ήρθαμε και σε επαφή με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι σε μία δοκιμή για τις μικρομεσαίες αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, να είναι ένα πρώτο βήμα. Η προσωρινή αξιολόγηση γίνεται, αλλά σε ποιο βαθμό αυτό δεν βρίσκεται στις ε, εκθέσεις. Και υπάρχει και μία διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι αξιολόγηση αυτές γίνονται Άρα λοιπόν η ποσοτικοποίηση πολλές φορές διαφέρει. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν λόγοι που οδηγούν σε αυτό. Μπορεί να μην βρίσκονται τα στοιχεία για να ποσοτικοποιήσει κανείς τα αποτελέσματα και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου οι ίδιες οι δοκιμές είναι και λίγο άσχετες με το αντικείμενο γιατί η νομοθεσία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το καλύτερο είναι να μην γίνει η δοκιμή. Υπάρχει πάντως χώρος βελτίωσης, γιατί όπως σας είπα έχουμε μεγάλες διαφεροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης οικονομικού αντίκτυπου. Από τις 22 εκθέσεις που μελετήσαμε, ε, καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν και κάποια παραδείγματα εναλλακτικών δυνατοτήτων για να επιτύχει στους πολιτικούς ε, στόχους. Δεν ξέρω αν οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίτηδε δεν εξετάζουν τα εναλλακτικά σενάρια. Κάποιε από τι ε, ενώσει επιχειρήσεων μα είπαν πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δει εναλλακτικέ δυνατότητε, αλλά δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα υπέρ η τη άποψη. Σε μόνο κάποιε περιπτώσει είδαμε να έχουν εξεταστεί και εναλλακτικέ λύσει ή να έχουν ε, προταθεί κάποια ελαφρεντικά μέτρα. Και τέλος, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό που βλέπουμε είναι να χρειάζεται βελτιωμένη ε, εξιολόγηση στις εκθέσεις οικονομικού αντίκτυπου. Αυτό θα μπορούσε γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έβλεπαν τότε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς δοκιμάζεται η νέα νομοθεσία που επηρεάζει τις μικρομεσαίες. Οι παρατηρήσεις μας λοιπόν ε, για το πώς χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πως οι κατευθυντές γραμμές επιτρέπουν μεγάλο περιθώριο διαφοροποίησης και θεωρούμε πως θα έπρεπε ε, να υπάρχουν περισσότερες, να είναι πιο συγκεκριμένες, να είναι πιο σφιχτές να καλύπτουν τι ανάγκε των υπηρεσιών και αυτό θα βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είχαμε μια καλύτερη παρουσίαση της δοκιμή στην ίδια την έκθεση. Δηλαδή να περιγράφουν το τι έκαναν, το τι δεν έκαναν, το πώς καταλήξαν σε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτό θα αποκάλυπτε το μυστήριο για το πώς τρέχουν αυτές οι δοκιμές. Θα πρέπει να παραδεχτούμε επίσης πως τρεχουν αυτες οι δοκιμε θα πρεπει να παραδεχτουμε επιση πω εχουμε και κάποιο πρόβλημα με την διαθεσιμότητα των στοιχείων σε κάποιες περιπτώσεις ε, δύσκολα λοιπόν βρίσκει κανείς ποιο είναι το ε, διοικητικό κόστος ε, για τις μικρομεσαίες αυτών των νέων προτάσεων. Η συστάση μας τέλος για τις ομάδες, για τους αρχάριους, είναι πως πρέπει να κάνουν κάποια πρώτα βασικά βήματα, να μην ασχολείται με αυτό μόνο μια ε, κυβερνητική υπηρεσία, αλλά ολόκληρη κυβέρνηση να αναγνωρίσει το ότι χρειάζεται πολιτική στο θέμα αυτό και σε κάθε περίπτωση να αξιολογείται η νέα νομοθεσία έτσι ώστε να γνωρίσουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο για τι μικρομεσαίε. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό βήμα. Να στηρίξουν τι δοκιμέ αυτέ και να είναι κάποιο υπεύθυνο, να υπάρχει μια αρμόδια, μια αρμόδια δομή κάποιος να λογοδοτεί έτσι ώστε να εξασφαλίσετε πως θα γίνονται οι δοκιμές. Αυτό είναι πολύ βασικό, αλλά είναι και κομβικό παράλληλα. Και τέλος θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε <coughs> αυτά τα εφαρμοστικά μέσα με κάποιους μετρήσιμους στόχους έτσι ώστε να προχωρήσουν να προχωρήσουν με την εφαρμογή. Για τη μεσαία ομάδα χρειάζονται συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Θα θέλαμε να παροτρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε αυτή την ομάδα να εγκρίνουν δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές, δεσμευτικές επαναλαμβάνω, και να συγκεκριμενοποιήσουν πώς θα πρέπει αυτές οι δοκιμές να γίνονται. Με ψηλά, να στοχεύουν ψηλά και στο πώς αξιολογούν τις ε, δοκιμές αυτές. Για τους προχωρημένους και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να προχωρήσετε και να δημιουργήσετε μια κουλτούρα καλύτερης ρύθμισης σε διάφορες κοινωνικέ υπηρεσίες με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας βοήθειας, ένα help desk, με την ε, διοργανική συνεργασία και βέβαια με κάποιους μηχανισμούς ανεξάρτητου ελέγχου όπως έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχει μια συγκεκρι... ένας φορέας ο οποίος αξιολογεί ε, και με τον τρόπο αυτό βελτιώνει ε, την εφαρμογή. Και θα πρέπει οι διάφοροι μεμονωμένοι κυβερνητικοί φορείς να βοηθηθούν στην εφαρμογή αυτών των δοκιμών. Αυτές είναι από τα, αυτά είναι κάποια από τα βήματα βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Να επιστρέψω τώρα στις συστάσεις. Όπως είπα και όταν ξεκίνησα, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της εφαρμογής Οπότε, εσείς θα πρέπει να επιφέρετε περισσότερη πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα εάν τα κράτη-μέλη έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά σε σε αν, σε άλλα, κάποια, σε άλλα κράτη-μέλη έχει υπάρξει, δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος, τότε θα πρέπει να υπάρξει έτσι ένας, να συμβαδίζουν στο ίδιο επίπεδο τα κράτη-μέλη μέσω αυτής της δοκιμής για τις μικρομεσαίες. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Το, η δοκιμή αυτή πρέπει να είναι ε, διαφανής και πρέπει να είναι ποσοδικοποιημένη και υποχρεωτική. Δεν νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει δοκιμή χωρίς αυτά τα βασικά στοιχεία. Πρέπει να ορίσετε στις κυβερνητικές υπηρεσίες πώς θα κάνουν το, τη δοκιμή και πρέπει να την παρακολουθήσετε κιόλας. Πρέπει επίσης να τη δείτε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσετε ε, για help desk και για δραστηριότητες κατάρτισης, ώστε να μπορούν αυτοί που θα ε, διεξάγουν την ε, δοκιμή όντως να την διεξάγουν σωστά. Κάποιος λοιπόν πρέπει να, έχει, να μπορεί να κάνει οικονομικούς υπολογισμούς των, υπολογισμούς των οικονομικών συνεπειών. Χρειάζεται λοιπόν και κατάρτιση για να υποστηριχτεί όλο αυτό. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να το ε, ενσωματώσετε σε μια γενικότερη προσέγγιση αξιολόγηση επιπτώσεων, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη νομοθεσία και η δοκιμή των ΜΜΕ είναι ένα, μια πτυχή του πώς βλέπουμε τη νέα νομοθεσία, ενσωματωμένη λοιπόν σε ένα πιο ευρύ σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων. take... ε, μπορώ λοιπόν να ολοκληρώσω εδώ την παρουσίασή μου. Αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαρίστω να απαντήσω. Ganz herzlichen Dank. Ευχαριστώ. Λεπτομερέστατη παρουσίαση. Ελπίζω να μπορέσετε εσείς να το διαβάσετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά, αλλά ευτυχώς που έχουμε τα έγγραφα. Ο κύριο Βέβερ έχει το λόγο, ο πρώτος. Παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη σχετικά με τη Γαλλία. Μιλήσατε για τις τρεις ομάδες, οι προχωρημένες, οι, ενδιάμεσες και οι αρχάροι, αυτοί που καθυστερήσαν, που καθυστερούν όμως δεν αναφερθήκατε στη Γαλλία, που είναι σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Γαλλία το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μία από τις αδυναμίες της γαλλικής οικονομίας, ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η αδυναμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα και εκεί, είναι, εκεί έγκυται η διαφορά ανάμεσα στην γαλλική αφενός και στη γερμανική, ιταλική και ισπανική οικονομία από την άλλη. Η πρακτική αυτών των δοκιμών ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι έχουμε αυτό το πρόβλημα των γαλλικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι σαφές ότι μια σειρά ε, νομοθετικών ρυθμίσεων αποτελούν και άλλη, άλλο, ε, άλλη μια δυσκολία για αυτές τις επιχειρήσεις. Επομένως θα ήθελα να ξέρω στη Γαλλία. Τι γίνεται με αυτές τις δοκιμές ε, των ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Χέρτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Πολύ αξιόλογα στοιχεία περιλαμβάνει. Θα ήθελα να ρωτήσω το πιο σημαντικό όμως που δεν το βρήκα μέσα σε αυτή την έκθεση. Είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό και την έκθεσή μου δεν τη γράψαμε για να ε, διευκολυνθούν απλώ ή να βελτιωθούν οι διαδικασίε. Τη γράψαμε έτσι ώστε οι μικρομεσαίε που είναι υπεύθυνε για το 1 τρίτο του ΑΕΠ και που είναι υπεύθυνε για το 2 τρίτα τη απασχόληση να έχουν καλύτερες δυνατότητες ώστε να μπορούν να προσθέσουν ε, κι άλλο. Ερώτημα λοιπόν, έχετε δεδομένα που να δείχνουν ότι σε αυτές τις χώρες που βρίσκονται στην, ε, στην προχωρημένη ομάδα οι μικρομεσαίες έχουν περισσότερα κέρδη και σε επίπεδο ΑΕΠ και σε επίπεδο απασχόλησης. Πώς θα περιγράφετε την προστιθέμενη αξία, Πού είναι η προστιθέμενη αυτή αξία. Είναι καλό να λέμε ότι ναι υπάρχει προστιθέμενη αξία, αλλά ποια είναι τελικά αυτή. Και εφόσον δεν μπορούμε να την καταστήσουμε προφανή αυτή την προστιθέμενη αξία, νομίζω ότι τελικά ένα, μια δοκιμή για τους δημοσίους υπαλλήλους κάνουμε αντί να προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις μηχανές για να μπορέσουν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχετε τέτοια δεδομένα. Αν δεν έχετε, έχετε σκοπό να τα βρείτε. Γιατί αυτό έχει την προστιθέμενη αξία. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσθέσουμε στο ΑΕΠ από την πλευρά των ΜΜΕ και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Οπότε, το ερώτημά μου είναι περισσότερο ο στόχος που έχουμε, γιατί το περιγράψατε κι εσείς. Εσείς περιγράψατε το μέσο. Εμένα όμως με ε, ενδιαφέρει περισσότερο ο σκοπός και όχι τα μέσα επίτευξή του, κυρίω για τις χώρες που βρίσκονται, δεν, βρίσκονται στο, δεν προχωρούν με το ίδιο βήμα με τις υπόλοιπε ε, χώρες. Ωραία, να σας δώσω το λόγο λοιπόν. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ο κύριος ε, Καλή θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα παρόμοιο ερώτημα. Υπάρχει σαφές οικονομικό όφελος στις χώρες που έχουν μπει στην ε, ομάδα των προχωρημένων και επίσης υπάρχει οικονομικό, οικονομική ζημία για τις χώρες που βρίσκονται στην ε, πιο ε, αρχική ομάδα. Είπατε, μιλήσατε για 23 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Το κόστος τελικά αυτής της ε, δοκιμής ποια είναι εάν εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και όχι μόνο σε αυτές που έχουν συμμετάσχει ήδη. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, συγγνώμη, κάτι ξέχασα. Ε, θα ήθελα να δω αν υπάρχει και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορών τομέων. Αν υπάρχει. Ή αν απλώς είναι το ίδιο για όλους τους τομείς. Γιατί εγώ θα θεωρούσα ότι κάποιοι ε, τομείς ε, θα ωφεληθούν περισσότερο από τη δοκιμή των ΜΜΕ από ό,τι άλλοι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σχετικά με το ερώτημα για το πώς η Γαλλία εφαρμόζει το, την δοκιμή ΜΜΕ, δεν κάναμε μια μελέτη συγκεκριμένα για την Γαλλία. Έχω απλώς τις γενικότερες απαντήσεις που έστειλε η Γαλλία στο ερωτηματολόγιο. Επομένως δεν μπορώ να, πω, να σας πω με λεπτομέρειες τι γίνεται. Έχω κάποια στοιχεία εδώ όμως που λέει ότι η δοκιμή του γίνεται ε, με συστηματικό τρόπο. Είναι μία από τις χώρες που εφαρμόζει ε, με τον πιο συστηματικό τρόπο την δοκιμή αυτή όταν ε, υπάρχει νέα νομοθεσία. Εκεί που χάνει η Γαλλία, αν θέλετε λίγο, είναι στην χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων. Και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για τη Γαλλία ε, για να δούμε κατά πόσον η Γαλλία χρησιμοποιεί λιγότερο προχωρημένες ε, μεθόδους. Θα επανέλθω, θα επανέλθω στην απάντηση αυτή μέσω της γραμματείας αφού εξετάσω τις απαντήσεις που μας έχει δώσει η Γαλλία. Τώρα, η... υπάρχει υψηλότερη ανάπτυξη στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ομάδα των προχωρημένων χωρών δεν τα είδαμε όμως αυτά όμως εμείς. Δεν είδαμε κατά πόσον ο τομέα αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πιο δυναμικός στις χώρες που εφήρμοσαν ε, πιο συστηματικά και με πιο προηγμένο τρόπο την, την δοκίμη. Δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση κατά πόσον το τεστ ε, είναι ένας λόγος για τον οποίο ε, αναπτύσσονται περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε δει αν, υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η δοκιμή μπορεί να αλλάξει την κατάσταση για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μια πολιτική θέση που λέει ότι ε, θα πρέπει υιοθετώντα μια νέα νομοθεσία θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει αυτή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη που θέλουν να τις εφαρμόσουν. Και στην ε, μελέτη που έγινε βλέπουμε ότι όντως ε, υπήρξε ε, αντίκτυπος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε, δεν έχουμε δει βέβαια τα δεδομένα, δεν έχουμε δει τα στοιχεία για το κατά πόσον υιοθέτησαν καλύτερη νομοθεσία, αλλά οι αξιωματούχοι μας είπαν ότι η δοκιμή έχει θετικές συνέπειες ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν εφαρμόσκονται στις γραμμές. Δηλαδή, επομένως, μπορεί να υπάρχει μπορεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην, ε, ε, στις επιδόσεις των, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην δοκιμή. Ελπίζω να απήντησα στην ερώτηση του κύριου Κέλλη. Αναφερθήκατε και στο κόστος εφαρμογής της δοκιμής. Εάν όντως θέλουμε να κάνουμε μια καλή δοκιμή, θα πρέπει να δαπανίσουμε και κάποιους πόρους. Και όντως υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, δεν έχουμε πόρους, ε, τα κράτη-μέλη δεν έχουν χρήματα, το ξέρουμε, όμως ε, χρειάζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ καλοί οικονομολόγοι για να γίνει σωστά η δοκιμή. Χρειάζεται δηλαδή μια ειδικευμένη ομάδα για να γίνει σωστά η δοκιμή. Ή μπορείτε να ζητήσετε και από την Κομισιό ε, να σας βοηθήσει. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τσάμπα, άρα κάποιο κόστος θα πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις για αν θέλουν να εφαρμόσουν τη δοκιμή. Αλλά με βάση τις απαντήσεις ε, που έχουμε, πιστεύουμε ότι θα είναι προ όφελο ε, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εν, γέννη, εάν ε, επενδύσουμε τους απαραίτητους πόρους για να ε, εφαρμόζει τη δοκιμή. Διότι αξίζει τον κόπο για να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης την έχουμε όλοι και γραπτός, μπορούμε να τη δούμε και με την ησυχία μας. Αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει, μπορεί να τη διαβάσει. Ευχαριστώ και για τα ερωτήματά σας. Μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό τη ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέτερσεν που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε για τώρα την ε, συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα.